can I invite all of you to take your chairs as soon as possible and as, as quiet and peacefully. Ε, καθίστε όσο πιο γρήγορα και όσο πιο ήσυχα γίνεται για να ξεκινήσουμε. I σας καλωσορίζω στην ε, συνεδρίαση λοιπόν της ε, Επιτροπής Αναφορών ε, και έχουμε και web streaming οπότε για όσους μας παρακολουθείτε από μακριά να σας πούμε ότι είναι η τελευταία μας συνεδρίαση πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα. Και βλέπω σήμερα εδώ πολλούς συναδέλφους παρόντες και βλέποντάς σας πραγματικά διαπιστώνω ότι όλοι έχουμε ανάγκη μία, ε, ένα παρατεταμένο θερινό διάλειμμα, γιατί πραγματικά η άνοιξη εδώ στις Βεξέλλες υπήρξε πολύ δύσκολη για μια σειρά από λόγους. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με την ε, συνεδρίαση. Ευχαριστώ την προσοχή σα στο σημείο 2 τη ημερήσια διάταξη, που είναι η έγκριση του σχεδίου ημερήσια διάταξη. Ε, σα παρακαλώ να λάβετε υπόψη σα το σημείο 29, η γνωμοδότηση σε ό,τι αφορά την πρόσβαση ε, στα φάρμακα και την οποία θα εξετάσουμε μετά το σημείο 11 τη ημερήσια διάταξη σήμερα. Ε, και να περνάμε στα πρακτικά της συνεδρίας της Δευτέρας Ιουνίου, ε, τα οποία έχουν διανεμηθεί. Αν δεν υπάρχουν ε, αντιρρήσεις, θεωρώ ότι εγκρίνονται και τα πρακτικά. Σας παρακαλώ να κάνετε ησυχία όσο γίνεται, γιατί πραγματικά είναι γεμάτη η αίθουσα ε, και δεν έχει καλή ακουστική, οπότε προσπαθήστε να ησυχάσετε λίγο και να με ακούτε λίγο πιο προσεκτικά για να έχουμε όλοι καλύτερη διάθεση. Να κάνω λοιπόν κάποιες ανακοινώσεις ε, από την πλευρά της Πρόεδρου. Ε, να σας πω ότι η γραμματεία θα αλλάξει ελαφρώς μετά από το καλοκαιρινό διάλειμμα και μεγάλη μου ικανοποίηση αλλά και με λίγο σας ε, ο, ο γιος Χερενές και ο γιος Γιωμούσα δύο δηλαδή πολύ έμπειρα ε, μέλη εδώ της ε, διοίκησης στο πλαίσιο και του συστήματος ε, κινητικότητας θα περάσουν στο Policy Department C που αυτό βέβαια για μας σημαίνει ότι θα χάσουμε δύο πολύ έμπειρα μέλη του προσωπικού μας, αλλά όχι για πάντα. Γιατί βέβαια το policy department αυτό το γάμα είναι και το δικό μας policy department οπότε θα μείνουμε σε επαφή και αυτό βέβαια είναι θετικό και ευχάριστο ότι δηλαδή θα σας χάσουμε έτσι, εντελώς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και τους δύο για τη δουλειά που κάνετε στη γραμματεία για μια σειρά από έτη και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο σαν νέα σας καθήκοντα και όπως είπα δεν θα είσαστε πολύ μακριά πότε θα σας βλέπουμε και ο Γιώργιο βέβαια θα συμμετάσχει και στην ε, ε, fact-finding αποστολή στο Ταράτο τον Νοέμβριο. Έτσι λοιπόν θα έχουμε δύο μέλη, νέα, ε, μετά από το θερινή διακοπή εργασιών, τα οποία θα συστήσω και κατά την πρώτη μας συνεδρίαση. Και υπάρχει και ένα μέλος το οποίο θα αποχωρήσει οριστικά από τη γραμματεία, ο Γιάρη Έρχολμ, καθώς συνταξιοδοτείται. Και με μπερδεύει λίγο αυτό δηλαδή αυτή η σύνταξη ενό τόσο ενό συναδέλφου. Οπότε συμμετέχει για τελευταία φορά ως ε, προσωπικό εδώ της Ένωσης ε, σε αυτή τη συνεδρία οπότε θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για όλα όσα έκανα και του εύχομαι κάθε επιτυχία όπου και αν βρεθεί, είτε στη Φιλανδία είτε στη Γαλλία, σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να, τον να χειροκροτήσουμε όλοι. συνάδελφοι. Ελπίζω τώρα να είναι παρόντες όλοι οι συνάδελφοι στην για να ψηφίσουμε και ελπίζω να έχετε όλοι μαζί σας και τις ε, κάρτες σας για την ψηφοφορία. So we will now vote on the mission report and recommendations. Ε, θα ε, ψηφίσουμε λοιπόν με του εγγράφου σε ό,τι αφορά τις συστάσεις μετά από την επίσκεψη στην Ισπανία. Έχουμε καταρχήν λοιπόν ε, τη συμβαστική τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σύσταση 1. Τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, όχι, καταπίπτει, καταπίπτει. Συγγνώμη, δεν ήμουν προσεκτική. Περνάμε στην τροπολογία 3. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίας αλλά ένα μέλο παραπάνω από την πλευρά του ΕΛΚΑ έχει ψηφίσει. Τώρα είμαστε εντάξει. Όχι, τώρα έχουμε ένα μέλο παραπάνω από του σοσιαλιστές. Τώρα είμαστε εντάξει. Πέρας λοιπόν τη ψηφοφορία και εγκρίνεται η τροπολογία. Περνάμε στην τροπολογία 4. Ψήφι πέρ. Κατά. Αποχές. Και εδώ θα πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. Δεν έχω ψηφίσει ακόμα όλοι. Τώρα λοιπόν. Είναι το πέρασμα της ψηφοφορίας και απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 5. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ τις 10 κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται α όχι να ελέγξουμε ηλεκτρονικά λοιπόν επί της τροπολογίας 11 ένα μέλος παραπάνω από το έλεγχο έχει ψηφίσει Πέρασε λοιπόν τώρα τη ψηφοφορία και απορρίπτεται η 11. Καταπίπτει. όχι, δεν καταπίπτει 12. Άρα ψηφίζουμε επί της 12. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να ελέγξουμε, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέρας λοιπόν της ψηφοφορίας και απορρίπτεται. Τροπολογία 13 ψήφι πέρα, Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. Πέρας. It has been approved. Amendment 17. Εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά Ας ψηφίσουμε, ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά, γιατί δεν ήταν σαφές. Επί της τροπολογίας 19 πάντα. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 20 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ελέγχουμε. Για την τροπολογία 22 λοιπόν, άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας, απορρίπτεται. 23 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να ελέγξουμε. Ηλεκτρονικά λοιπόν για την 27 ψηφίζουμε. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 28 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Α, όχι, καταπίπτει, συγγνώμη, 30. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 36 καταπίπτει γιατί εγκρίθηκε 35 οπότε ψηφίζουμε επί του συνόλου του εγγράφου. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. And Πέραση της ψηφοφορίας εγκρίνεται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 Επόμενο θέμα, το πιλωτικό πρόγραμμα για το bullying. Και πάλι, ενιαία ψηφοφορία. Μπορούμε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, μάλλον άπαξ, έναρξη ψηφοφορίας. It's a single vote. The vote is still open and now it's closed. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται Σε Συγχαρητήρια στη Σολεδάδη. Ας περάσουμε τώρα στα σημεία των αναφόρων. Παρακαλώ όσοι αποχωρείτε να το κάνετε όσο γίνεται πιο ησυχά.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 Όσοι δεν θέλουν να παραμείνουν για τις αναφορές, παρακαλώ αποχωρήστε ησύχως όσο γίνεται πιο σύντομα. So the next item that we will το επόμενο σημείο που θα εξετάσουμε είναι η αίτηση 709 του 2015 του Χάνες Βίλεμ Κέλ για την προστασία της πολιτισμικής ταυτότητας και την επιβίωση της ε, κοινότητας των Σόρβων. Παρίσταται ο αναφέρον, κύριος Κέλ. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά, παρακαλώ. Δυστυχώ δεν είναι όλοι εξίσου ευγενεί. Του έχω ζητήσει πολλάκι να αποχωρήσουν από την αίθουσα και δεν το κάνουν. So now I am happy to invite you to take the Ωραία, έχετε το λόγο λοιπόν για πέντε λεπτά για την αναφορά σας. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte die Gelegenheit... Αξιότιμοι κύριε και κύριοι, θα ήθελα εδώ να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να σα συνοψίσω τα κύρια σημεία αυτής τη αναφοράς και σα ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Εγώ εκπροσωπώ ως εκπρόσωπος της ε, ε Συμμαχίας ε, των Σόρβων, ακριβώς αυτή την εθνική ομάδα των ε, Σόρβων και αποτελούμε ως οργάνωση την πολιτική πλατφόρμα των για την προάσπιση των συμφερόντων των Σόρβων και εκπροσωπούμε γύρω στους 120.000 Σόρβους δηλαδή γύρω στο 90% της, των κατοίκων εκεί. καταρχήν τίθεται ένα ερώτημα εδώ σε ό,τι αφορά την αναφορά μας ε, ε ως προς την εφαρμογή του εθνικού σε σύγκριση με το νοσιακό δίκαιο. Ε, από την άλλη πλευρά ε, θέλουμε να εφαρμοστεί να εφαρμοστούν οι διατάξεις που έχουν κατοχυρωθεί στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σε ό,τι αφορά την προστασία των ε, θύμων και των παραδόσεων των ε, μικρότερων κοινοτήτων. Ε, προφανώς η διατήρηση αυτών των θύμων και της γλώσσας των τσόπων εξαρτάται και από τη διατήρηση του περιβάλλοντος στην περιοχή στην οποία κατοικούν. 136 χωριά χάθηκαν στην ευρύτερη περιοχή των Σόρμπων, καθώ χρειάστηκε να μετεγκατασταθούν και ακόμα 12 χωριά προβλέπεται πω θα μετεγκατασταθούν λόγω ακριβώ τη δημιουργία ηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ενέργειας από Και πάντοτε βέβαια ε, με αυτές τις μετακαταστάσεις χάνονται τα πάντα. Δηλαδή χάνεται όλη η κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική ταυτότητα της ευρύτερης ε, περιοχής. Ε, και εμείς διαπιστώνουμε ότι βάσει τις αιτήσει που έχουν υποβληθεί τίθεται σε κίνδυνο ακόμα 7 χωριά. Και εμείς σας καλούμε λοιπόν να προβείται νομικά κατά αυτών των ενεργειών οι οποίες ουσιαστικά παραβιάζουν την νομοθεσία ε, που υφίσταται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, προστασία των σχετικών ε, μειονοτήτων. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρξει μια προστασία του σχετικού Ε, προστασία των, ε, των ε, σχετικών κοινοτήτων και με βάση την εφαρμογή του άρθρου 160 της ΑΕΛΟ και από εκεί και μετά. Ως δεύτερο σημείο, προφανώς οι εξωτερικές δραστηριότητες σε αυτό το τομέα δεν αποτελούν αντικείμενο το οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο όμως η μόλυνση του υδρόβιου ορίζοντα των επιφανειακών οδάτων της ατμόσφαιρας είναι ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της. Και στο Λάος πραγματικά υπάρχει συνεχής επιμόλυνση με βαρέα μέταλλα, με οξύδια του θείου ε, των υδάτων και ε, στην ε, δική μας αναφορά αναφέρεται μία ακόμα, ένας ακόμα σε κίνδυνος, ότι δηλαδή προβλέπεται μία δημιουργία ενός ακόμα μιας ακόμα εξωτικής περιοχής στα σύνορα του Λάουζιτ και βέβαια ακριβώς επειδή πρόκειται για παρόμοια δραστηριότητα με αυτές που λαμβάνουν ήδη η χώρα θα έχουμε αντίστοιχε ε, ε, μολύνσει. Και βέβαια αντίστοιχε περιπτώσει είχαμε και στο παρελθόν, όπου είδαμε δηλαδή ποια ήταν η μόλυνση από την ε, παγωγένεια με βάση των ε, το λίγο. Οι σχετικέ πληροφορίε είναι διαθέσιμε ε, σε διάφορες χώρες τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί, λοιπόν θα θέλαμε να ξεκινήσει μια δικασία κατά παράβαση εναντίον τη Πολωνία, ε, προκειμένου να διασφαλίσουμε την προστασία του περιβάλλοντος ειδικότερα των υδάτων και της ατμόσφαιρας στην περιοχή τη Πολωνίας θα θέλαμε να ξεκινήσει μια, ή να ναι. ληφθεί πιο σοβαρά αυτή η διετή έκθεση η οποία ε, υποβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται από εδώ ε, και πέρα και ζητήματα τέτοια περιβαλλοντική προστασία και παραβιάσεων τη νομοθεσία. Ένα ακόμα σημείο είναι ότι προφανώς αποτελεί η εξωτερική βιομηχανία ε, εθνικό δικαίωμα, αλλά από την άλλη πλευρά οι κατευθυντήρες γραμμές σε ό,τι αφορά τους στόχους για την ε, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ε, και της προστασίας του περιβάλλοντος θα πρέπει να τύχουν σε βασμό. Αυτές, αυτές λοιπόν οι παραβιάσεις εναντίον τέτοιων λαμβάνουν χώρα στο Λάουζιτς θεωρούμε πως ε, με την ε, περαιτέρω επέκταση της, ε, των εξορίξεων σε αυτή την περιοχή και με την, με την περαιτέρω δημιουργία σταθμών παραγωγής ενέργειας θα, θα πολλαπλασιαστούν ακόμα περισσότερα τα προβλήματα. Και βέβαια η, η εξόριξη λύνεται στην ευρύτερη περιοχή ενισχύεται και κρατικά, με αποτέλεσμα βέβαια να εντατικοποιούνται αυτές οι δραστηριότητες και να είναι απαραίτητο στη συνέχεια να χρειαστούν κάποια, ε, να ληφθούν κάποια μέτρα εξυγίανσης στο ευρύτερου περιβαλλόντος. Ε, ε, με αυτόν τον τρόπο βέβαια με ε, αυτές τις κρατικές ενισχύσεις δεν διασφαλίζεται και ο υγιής ανταγωνισμός εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας καλούμε λοιπόν να διασφαλίσετε ότι δεν υπάρχει παράβαση των σχετικών διατάξεων και τη Συμφωνίας για την Προστασία του Περιβάλλοντος και στο πλαίσιο της COP21 από την πλευρά της Πολωνίας. Η οι παραβιάσεις οι οποίες αφορούν την εθνική νομοθεσία σε ό,τι αφορά την προστασία των αγρίων ειδών ε, είναι ένα ακόμα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Έχουμε δει ότι στην ευρύτερη περιοχή έχουν καταστραφεί μία σειρά από είδη πανίδα και χλωρίδας και οι διατάξει, οι οποίε προβλέπουν την εφαρμογή των σχετικών ε, οδηγιών δεν εφαρμόζονται και δεν υπάρχει σεβασμό από την πλευρά των αρμόδιων αρχών. Πολλά δηλαδή είδη τη ε, χλωρίδα και πανίδα δεν ε, συνεχίζουν να απειλούνται με εξαφάνιση ή έχουν εξαφανιστεί από την ευρύτερη περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα πρέπει να ξε... μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία κατά παράβαση κατά αυτών των αρχών ακριβώς ε, επειδή θα πρέπει να διασφαλιστεί η κατάλληλη προστασία των ε, ειδών. Ε, σας ευχαριστώ για μία ακόμα φορά θερμά για την υποστήριξή σας. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Πρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχω τρία ονόματα. Όποιος θέλει, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον αναφέροντα για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή παρουσίαση. Δεν χρειάζεται να συνοψίσουμε και πάλι την αναφορά. Θα εστιάσω στα κύρια σημεία. Πρώτον, να τονίσω ότι εξετάσαμε μεγάλη προσοχή την αναφορά και έχουν ε, συμμετάσχει στην ανάλυση και εξέταση ε, πολλές ε, γενικές διευθύνσεις, δικαιοσύνης, ενέργειας, περιβάλλοντος, καθώς και Γενική Διεύθυνση Παιδείας και Πολιτισμού και Ανταγωνισμού. Η Γενική Διεύθυνση από τη Δικαιοσύνη και από το Περιβάλλον είναι μαζί μου σήμερα για να απαντήσουν ε, σε τυχόν ερωτήσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα τις συγκεκριμένες εκκλήσεις ε, του αναφέροντα, εντοπίζουμε τρία κύρια μηνύματα. Στήριξη για την ε, διατήρηση του πολιτισμού και γλώσσας των Σόρβων. Δεύτερον, να εξετάσουμε τι θα γίνει με το μέλλον της εξόριξης άνθρακα και τη χρήση του σε όλη την Ευρώπη και τρίτον συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες σχετικά με την ποιότητα των υδάτων και της ατμόσφαιρας. Θα εξετάζουμε τη σειρά. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, πρέπει να τονίσουμε ότι οι διακρίσεις με βάση τη συμμετοχή σε μία ε, μειονότητα απαγορεύεται αυστηρά από την ε, Χάρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν το κοινοτικό δίκαιο, ε, δεν ε, μπορούμε εμείς να επισέλθουμε σε όλο αυτό ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το μοναδικό θεσμικό όργανο το οποίο μπορεί να παρέμφει είναι η χάρτα του Συμβουλίου του της Ευρώπης για τα δικαιώματα των μειονοτήτων που έχει κυρωθεί και από τη Γερμανία. Επομένω, οι εξουσίε ε, τη Επιτροπή, σε ό,τι αφορά την αναγνώριση του καθεστώτος μειονοτήτων είναι ε, περιορισμένε, όμως έχουμε προγράμματα όπω είναι το Erasmus Plus και έτσι ομάδες ε, και κοινότητε που προσπαθούν να υπερασπιστούν δικαιώματα μειονοτήτων μπορούν να κινηθούν αρκεί να καταδεικνύονται ορισμένε προποθέσει. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σημείο, για το μέλλον της εξόριξης άνθρακα και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην περιφέρεια και ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε ότι η χρήση άνθρακα μειώνεται σε ό,τι αφορά το ενεργειακό μείγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τις τελευταίες δεκαετίες αυτή είναι η τάση και θεωρούμε ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον και στη Γερμανία. Ταυτόχρονα, πρέπει να τηρήσουμε και το άρθρο 194 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να προσδιορίσουν τις ε, συνθήκες για την αξιοποίηση των ενεργειακών τους πόρων, μπορούν να καθορίσουν το ενεργειακό τους μείγμα και την γενική δομή της, ε, παροχής ενέργειας. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, έχει την αρμοδιότητα να απαγορεύσει ε, την εξόριξη άνθρακα ή να καταργήσει σταδιακά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνθρακα, παρότι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει μια σταδιακή τάση μείωσης αυτού του φαινομένου. Τρίτο θέμα που τόνισε ο αναφέρον στην παρουσίασή του είναι η επιβολή της συμμόρφωσης με τους ευρωπαϊκούς κανόνες σε ό,τι αφορά την ποιότητα των υδάτων και της ατμόσφαιρας. Για την ε, ατμόσφαιρα έχουμε δύο νομοθετικές πράξεις, ε, οδηγία περί βιομηχανικών εκπομπών και οδηγία για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Η Επιτροπή έχει εξετάσει τι ισχύει ε, για τη συμμόρφωση στη Γερμανία με αυτές τις δύο νομοθετικές πράξεις. Για την πρώτη οδηγία βιομηχανικών εκπομπών όλα τα Όλε όλες οι μονάδες παραγωγής ενέργεια άνω το 50 ΜΒ στη Γερμανία θα πρέπει να ε, εφαρμόζουν ε, τις βέλτιστες ε, δυνατέ τεχνικές και από ό,τι βλέπουμε δεν υπάρχει παράβαση αυτών των κανόνων και σε ό,τι αφορά την οδηγία περί ποιότητας της ατμόσφαιρας παρότι δεν υπάρχει παράβαση των ευρωπαϊκών κανόνων οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν εντοπίσει παραβάσεις σε γειτονικές περιοχές. Πρέπει λοιπόν να κινηθούν διαδικασίες, έχουν ήδη ξεκινήσει μάλλον νομικές διαδικασίες για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων ε, στη Γερμανία, στην Πολωνία και στην Τσεχία. Θα μείνω εδώ. Όπω είπα, έχουμε και συναδέλφους από την Γενική Διεύθυνση δικαιοσύνη, και Περιβάλλοντος για να απαντήσουν αν υπάρχουν πιο συγκεκριμένα εξειδικευμένα ερωτήματα. Σας ευχαριστώ πολύ, πρόεδρο και τους δύο, αλλά και, τον, και σας και τον αναφέροντα για την ε, πολύ καλή αυτή αναφορά και ακριβή απάντηση. Το λόγο ε, τώρα έχουν οι συνάδελφοι. Ήδη κυρία Στανόκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Έχω δει με τα μάτια μου την περιοχή αυτή. Το Πήγαμε πριν από ένα χρόνο. Είχαμε εκεί τη συνδιάσκευση ε, του αδερφού κόμματός μας. Με εκπλήσει ιδιαίτερως η εκτίμηση της Επιτροπής ότι δεν υπάρχει καμία παράβαση ε, της ε, οδηγίας περί υδάτων ε, του προγράμματος του Natura 2000 και της ποιότητας της ατμόσφαιρας. Γιατί το είδαμε τα ίδια μας τα μάτια. Πώς γίνεται αυτό. Ακούσαμε τον αναφέροντα. Μόλις εγκρίναμε μία έκθεση για την διαρευνητική μας αποστολή σε δύο ποταμούς στην Ισπανία. Πρόπερση πήγαμε στη Γαλλικία. Επομένω, είδαμε με τα ίδια μάτια και τη ρήπανση, την πολύ άσχημη κατάσταση για τους ε, κατοίκους της περιοχής και τώρα οι εμπειρογνώμονες τι λένε όλα βαίνουν καλώς. Μα πώς είναι δυνατόν. Αυτό είναι το ερώτημά μου προς ε, την Επιτροπή, γιατί είπατε ότι δεν ήσασταν ακριβώ εκείνη την περιοχή, πήγατε σε γειτονικέ, ε, στην Τσεχία. Από πού προκύπτει λοιπόν αυτή η πραγματογνωμοσύνη. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, Και εγώ είχα πει να αναφέροντα να υποβάλει αυτή την αναφορά. Τα έχω δει λοιπόν. Δυστυχώς δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στη σύμβαση. Σε τη φορά ακόμα και την επέκταση της εξόριξης άνθρακα. Η Γερμανία με την κατάργηση των ε, εργοστασίων πυρηνική ενέργειας χρησιμοποιεί μεγαλύτερε ποσότητες άνθρακα και υπάρχουν ακόμα και ανησυχίες για επέκταση αυτής της περιοχής εξόριξης και βλέπουμε στα χωριά που ζουν οι σόρβοι και τώρα περνάμε στην άλλη πλευρά της υπόθεσης, τη διατήρηση δηλαδή της παράδοσης και της παραδοσιακής περιοχής αυτής της μειονότητας. Η Επιτροπή μας ε, παραπέμπει στην Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, αναφέρει μειονότητες και συγκεκριμένα γλωσσικές μειονότητες. Εσείς απαντάτε ότι δεν είναι δεσμευτικά όλα αυτά και δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Ξέρουμε ότι τα πράγματα χειροτέρεψαν μετά την πώληση του ορυχείου. Η Waterfall ήταν ε, ε, η προηγούμενη κάτοχος, μια σουηδική επιχείρηση, τώρα πωλήθηκε σε μια τσεχική εταιρεία που μπορεί να επεκτείνει αυτές τις δραστηριότητες. και εκπροσωπώ εδώ και την συνάδελφο Βάλερο από το Σουηδία, την οποία ενδιαφέρουν ιδιαίτερως σε αυτά τα ζητήματα. Όμως δυστυχώς ε, είναι σε μία αποστολή της ΛΥΜΠΕ στο Καλέ. Όμως ε, παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή την υπόθεση. Παρακαλώ κύριο Σεβαστιά, σας παρακαλώ να μην επαναλαμβάνετε τα ίδια και να είστε ακριβείς. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ είδα με τα ίδια μου τα μάτια τα όσα συμβαίνουν στην ε, περιφέρεια στην οποία ε, ε, ζουν οι Σόρβοι. Είδαμε κατάφορη παραβίαση του ε, ευρωπαϊκού πνεύματος ε, και των κανόνων που το πνεύμα αυτό διέπουν. Ε, επίσης, από την άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι δεν έχουμε καμία, κανένα σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και όχι μόνο δεν τους δίνουν σχολεία για να μαθαίνουν τη γλώσσα τους και να τη διδάσκονται, αλλά τους δημιουργούν και προβλήματα με το περιβάλλον. Εγώ επανέρχομαι στο πρώτο θέμα. Ε, βάσει των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αξιών της ε, θα πρέπει τα παιδιά των σόβρων να έχουν τη δυνατότητα να διδάσκονται στη γλώσσα τους. Μιλάμε εδώ για μια περιοχή η οποία είναι πάρα πολύ ευαίσθητη και η οποία ε, παραβιάζεται ε, ε, και της οποίας μάλλον τα δικαιώματα παραβιάζονται όσον αφορά και τα δικαιώματα στη διδασκαλία και όσον αφορά τα δικαιώματα που έχουν στο περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθορίσει κάποιες στρατηγικές όπως ας πούμε η 2020 και επίσης έχει προσυπογράψει για τις συμφωνίες της COP21 στο Παρίσι έτσι ώστε να μπορέσει να εναρμονίσει την παραγωγή και την ενέργεια και το περιβάλλον. Ε, και διαπιστώνουμε εδώ, ενώ η Γερμανία γενικώ συμβαδίζει με τις αρχές αυτές, τα ειδικά στοιχεία τούτης εδώ της περιοχής, τούτης εδώ της περιοχής αντιτίθενται στο γενικό ε, προγραμματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μέλλον. Τρίτον, ε, εκπλήσωμε όπως και η συνάδελφος Ζανόκα, που η εκπρόσωπος ε, της Κομισιόν δεν βλέπει καμία παραβίαση των, της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος και του υδροφόρου ορίζοντα. Είναι... Πώς είναι δυνατόν να μας λέει ότι είναι τόσο σαφές ότι δεν υπάρχει ε, καμία παραβίαση όταν εμείς έχουμε δει με τα ίδια μας τα μάτια την κατάσταση και έχουμε διαπιστώσει την ε, ε, καταστροφή του περιβάλλοντος και άλλωστε είναι προφανές ότι όλα τα ανοιχτά ορυχεία αποτελούν μεγάλο πρόβλημα για το περιβάλλον. Νομίζω ότι θα πρέπει να στηρίξουμε τους αναφέροντες είναι, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η βαρύτητα όλων των ε, στοιχείων εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλη και όσον αφορά την ε, μόλυνση και όσον αφορά τη μη προστασία του περιβάλλοντος και όσον αφορά τη μη παροχή διδασκαλίας και άλλων δικαιωμάτων σε, αυτούς, τους, ε, σε αυτό το λαό των Σόρβων και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να στείλουμε αποστολή εκεί και να προωθήσουμε το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κάμπρας. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Βρέθηκα και εγώ σε αυτή την περιοχή και δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα ήδη υπόθηκαν. Απλώς θα ήθελα πολύ σύντομα να πω ότι συμφωνώ με τα όσα υπόθηκαν από πλευρά του αναφέροντα και ότι υποστηρίζω πλήρως τα όσα είπε σε ό,τι αφορά τις ε, τρεις ε, πτυχές τις οποίες έθιξε. Πρώτον, θα πρέπει πράγματι να προστατεύσουμε και να υποστηρίξουμε ε, την γλώσσα και τα έθιμα της σοβικής κοινότητας. Δεύτερον, πράγματι θα υπάρξουν ε, τρομακτικές συνέπειε σε περιβαλλοντικό επίπεδο λόγω των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στην ε, περιοχή. Και θα ήθελα επίσης να πω ότι υποστηρίζω την έραξη μια διαδικασία κατά παράβαση τόσο εναντίον τη Γερμανία όσο και εναντίον τη ε, Πολωνία ε, σε ό,τι αφορά την χρήση του λιγνίτη και επαναλαμβάνω ότι ε, υποστηρίζω 100% ε, το αίτημα αυτό του πληθυσμού ε, της περιοχής των Σόρων. Ευχαριστώ. Είναι περίπλοκη αυτή η αναφορά, γιατί θίγει πολλά και διαφορετικά ζητήματα. Θα ήθελα τώρα να στραφώ και πάλι στον αναφέροντα για δύο λεπτά. Εάν έχει κάποιες καταληπτικές παρατηρήσεις, αν θέλετε κάτι να προσθέσετε στα όσα υπόθηκαν τώρα που ακούσαμε και τα μέλη της Επιτροπής. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά και μετά θα προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, συμπληρώνοντας ε, με βάση τα όσα ακούσαμε και τώρα από την Επιτροπή, να πω ότι οι εξορρυκτικές δραστηριότητες ε, αποτελούν ε, το βασικό πρόβλημα για όλα τα προβλήματα που έχουν προκύψει στην περιοχή. Οπότε εκείνο που έχει αποφασιστική σημασία είναι το κατά πόσο μπορούμε να στραφούμε ενάντια ε, σε αυτήν την εξορρυκτική βιομηχανία η οποία εμπίπτει ακριβώς στις εθνικές αρμοδιότητες ή εάν θα πρέπει να εστιάσουμε στι περιβαλλοντικέ ε, επιπτώσει, ε, και κατά αυτόν τον τρόπο βέβαια θα μπορούσαμε να επηρεάσουμε την εξωτερική βιομηχανία και τι δραστηριότητε. εκεί. Νομίζω πω αυτό είναι ο ενδεδειγμένος ε, τρόπο, και σα ευχαριστώ όλου για την υποστήριξή σα. Λοιπόν, προτείνω βεβαίω να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και θα ήθελα κύριε Κέλ να σα ενθαρρύνω να στραφείτε στο συνήγορο του πολίτη στη Γερμανία ναι, υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχει συνήγορο του πολίτη στο δικό σα κρατήδιο, στον οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε και στη σχετική Επιτροπή Αναφορών. Γιατί πολλά από αυτά τα ζητήματα είναι θέματα εθνική αρμοδιότητας. Αυτό είναι το πρώτο λοιπόν. Να απευθυνθείτε στην Επιτροπή Αναφορών στο κρατήδιό σας. Θα ε, προσπαθήσετε να βρείτε λοιπόν τον συνήγορο του πολίτη στην περιοχή σας για αυτά τα ζητήματα εθνικής αρμοδιότητας, όπως ο καθορισμός του ενεργειακού μείγματος. Αυτό είναι θέμα εθνικής αρμοδιότητας. Επίσης, κύριε Κέλ, σας παροτρύνω να δώσετε και στη δική μας Επιτροπή περισσότερες πληροφορίες σε ό,τι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για ε, τον καθαρισμό των αποβλήτων από την εξαιρετική βιομηχανία. Αν μπορείτε να το κάνετε αυτό εντός δύο μηνών θα ήταν εξαιρετικό. Και όταν θα έχουμε αυτές τις ε, πληροφορίες θα θέλαμε να στραφούμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξετάσει αυτά τα νέα στοιχεία που θα μας δώσει ο αναφέρον και να υπάρξει συνέχεια. Προτείνω επίσης να αποστείλουμε επιστολή ε, στα κρατηδία της Αξονίας και του Βρεδεμβούργου και εκεί να εκφράσουμε τον προβληματισμό μας για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και να ζητήσουμε και από εκείνους ε, πληροφορίες για συγκεκριμένα περιβαλλοντικά ζητήματα που έθιξε ο αναφέρον. Και αυτό είναι προς το συμφέρον και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι κάτι που ενδιαφέρει δηλαδή τέλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στις συνθήκες και στη χάρτα για την ε, διατήρηση των μειονοτήτων, της γλώσσας και του πολιτισμού είναι κάτι μη αμεληταίο. Πρέπει να τα διαφυλάξουμε όλα αυτά και να υπογραμμίσουμε ότι είναι ζητήματα πολύ σημαντικά για την Επιτροπή μας και για το Κοινοβούλιο εν γέννη. Επομένω, ε, θα αποστείλουμε επιστολή ακριβώ για αυτό το ζήτημα, η Μάργαρετ. Συμφωνώ απολύτω και νομίζω ότι η Επιτροπή κάνει ό,τι μπορεί για να ξεφορτωθεί αυτή την υπόθεση. αντί να μελετήσει σε βάθος. Ακόμα και δεν μπορεί να κινηθεί η διαδικασία επί παραβάση. Παραμένει δική μας ευθύνη να εξετάσουμε αυτές τις καταγγελίες πολιτών για πιθανόν πολύ σημαντικές ε, παραβάσεις της Ευρωπαϊκής Αμαθησίας για την ε, ατμόσφαιρα, για τα ύδατα και το καθεξής. Επομένως, πρέπει να το πάμε πολύ στα σοβαρά, ακόμα και αν δεν μπορούμε να κινήσουμε διαδικασία παραβάση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό θέμα για τα μέλη αυτής της Επιτροπής γιατί είναι μια πολύ ανησυχητική κατάσταση από ό,τι βλέπω. Από την απάντηση της Κομισιόν ε, γνωρίζουμε ότι ήδη υπάρχει δικασία παραβάση κατά της Γερμανίας ό,τι αφορά την, ατμόσφαιρα, τη ρήπαση της ατμόσφαιρας. Όμως δεν συμπεριλαμβάνει αυτή την περιοχή. Όταν λάβουμε περαιτέρω στοιχεία θα το εξετάσουμε περαιτέρω και η Επιτροπή βεβαίω ε, και θα το μελετήσουμε σε βάθος. Όμω ένα σύντομο κείμενο, υπάρχουν τόσα ζητήματα σημαντικού ενδιαφέροντος. Συμφωνούν οι συνάδελφοι με την πρότασή μου. Ωραία. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και εσάς κύριε Κέλ που ήρθατε μέχρι εδώ και μας κάνετε αυτή την παρουσίαση. Να θυμάστε ότι αυτά απασχολούν ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο εσάς. Ωραία, επόμενη αναφορά 0603 ε, για ένα εργοστάσιο παραγωγής και στο Βαγιαδολίδ. Ο κύριος Μιλάγρος Μάρκος Ορτέγα είναι εδώ και εκπροσωπεί τον αναφέροντα. Καλώς ήρθατε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά και μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση. Buenos días, señoras y señores diputados. Vengo... Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έρχομαι εδώ σε αυτήν την συνεδρίαση διότι είμαι σύμβουλος γεωργίας και κτηνοτροφίας της περιφερειακής κυβέρνησης, της αυτόνομης κυβέρνησης της Καστίγια Ελαιών και συγκεκριμένα υπεύθυνη για την γεωργική πολιτική, την πολιτική διατροφής εκπροσωπώντας εδώ ε, και το Σωματείο για την διατήρηση των επιχειρήσεων ε, στην Καστίγια Ελαιών. Ε, εμείς σαν οντότητα είμαστε υπεύθυνοι για τις διαδικασίες ε, ε, κρίσεων των ε, επιχειρήσεων και συμμετέχουμε ενεργά σε όλες τις διαδικασίες της διακυβέρνησης. Πρέπει να σας πω ότι δύο μήνες πριν ε, την ε, ανακοινωθήσα πάυση των εργασιών ε, που θα οδηγήσει στο κλείσιμο της, του εργοστασίου και στην ανεργία 85 κτηνοτρόφους, 85 εργαζόμενους αλλά και πάρα πολλούς κτηνοτρόφους οι οποίοι δίνουν το γάλα τους ε, κάθε μέρα ε, σε αυτό το ε, εργοστάσιο είναι εξαιρετικά επίκαιρη η συζήτηση. Η τοπική κυβέρνηση αλλά και όλη η δημόσια διοίκηση ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το θέμα αυτό. Έχουν γίνει πάρα πολλές συνεδριάσεις με τα υψηλόβαθμα στελέχη αυτής της εταιρεία, αλλά χωρίς αποτέλεσμα ακόμα και η Ισπανική πρεσβεία στην Γαλλία συμμετείχε στην διαδικασία αλλά χωρίς αποτέλεσμα πάντα. Ε, όλα αυτά οδηγούν εν τέλει στο κλείσιμο και την πάυση δραστηριοτήτων αυτής, της, ε, αυτού του εργοστασίου στο Βαγιαδολίθ. Ε, δυστυχώς δεν καταφέραμε μέχρι τώρα να αλλάξουμε την γνώμη των ηθινόντων αυτής της επιχείρησης και αυτού του εργοστασίου. Ε, δεν είναι η πρώτη φορά, δεν είναι η πρώτη αλλά ούτε και η τελευταία ε, περίπτωση κλεισίματος δραστηριότητας. Ε, όμως δεν μας οδηγεί αυτό σε ενώπιον της Επιτροπής σας. Εμείς έχουμε έρθει εδώ γιατί θεωρούμε ότι το θέμα αντιτίθεται σε βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την συνοχή, όσον αφορά την κοινωνική ευθύνη και όσον αφορά και τον ανταγωνισμό. Για πρώτη φορά βλέπουμε σημαντική παράβαση, παραβίαση παραβίαση των ε, δικαιωμάτων των εργαζομένων διότι ε, ε, προχωρεί μια επιχείρηση σε προαναγγελθήσα και αδικαιολόγητη πάυση των δραστηριοτήτων. Μέχρι τώρα είδαμε ε, ότι ε, η παραγωγή αλλά και η χρήση ε, του εργοστασίου έχει πέσει στο 50%. Αυτό δεν είναι αποτέλεσμα προβλημάτων αλλά είναι αποτέλεσμα ενός προσχεδιασμένου σχεδίου το βάση του οποίου μεταφέρεται εξοπλισμός και δυνατότητα από αυτό το εργοστάσιο σε άλλες. Ε, ε, επίσης ε, πρέπει να σας πω ότι ακόμα και με το 50% της παραγωγής τους η εταιρεία έφτασε να έχει 2 εκατομμύρια ευρώ τζίρο στο τελευταίο, στο τελευταίο, στην τελευταία χρήση. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, κατά δεύτερο λόγο θα ήθελα να θίξω το θέμα της χρήσης πόρων από το, από τα διαφορετικά ευρωπαϊκά ταμεία. Ε, χρησιμοποιήθηκαν τα χρήματα αυτά με τον στόχο να ε, ενδυναμωθεί η παραγωγή της ίδιας αυτής εταιρείας, ε, της ίδιας αυτής επιχείρησης σε, άλλες, σε άλλα εργοστάσια. Αυτά τα χρήματα λοιπόν, τα οποία βοήθησαν την ανάπτυξη άλλων εργοστασίων, ε, τώρα δίνουν την δυνατότητα σε αυτήν την επιχείρηση να κλείσει τον λόγο εργοστάσιο και να μεταφέρει την δραστηριότητά της σε άλλο. Ε, ο στόχος των διαρθρωτικών ταμείων όμως, από όσο γνωρίζουμε, είναι ε, να ε, καλυφθούν τα μειονεκτήματα ορισμένων περιοχών και να επέλθει μια ισορροπία όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Με κανένα τρόπο δεν θέλουν νομίζω τα διαρθρωτικά ταμεία να αναπτύξουν κάποιες περιοχές ή κάποια εργοστάσια προς ζημίαν άλλων και να οδηγήσουν σε κλείσιμο κάποιων άλλων εργοστασίων. Ακόμα περισσότερο όταν η επιχείρηση στην οποία δόθηκαν τα χρήματα αυτά ε, δεν ε, επιτρέπει αυτή η, ε, αυτό το εργοστάσιο να αγοραστεί εν τέλει από κάποιον άλλον παραγωγό έτσι ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί η διαδικασία. Γιατί θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει ανταγωνισμός απέναντί της. Φτάνω στο τελευταίο σημείο. Θεωρούμε ότι εδώ έχουμε παραβίαση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έτσι όπως αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζουμε ότι η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων είναι βεβαίως μια εθελοντική διαδικασία, αλλά αυτή η προσχεδιασμένη και αδικαιολόγητη μετάθεση των, ε, του εργο, των δραστηριοτήτων του εργοστασίου Ιντούστριας Λάκτεας ε, ε, είναι μια πάρα ένα πάρα πολύ ισχυρό χτύπημα ε, στις ε, αρχές τις οποίες, οι οποίες θα πρέπει να διέπουν το επιχειρήνι στην Ευρώπη. Δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα σε 85 οικογένειες και γι' αυτό στραφήκαμε σε εσά. Ευχαριστώ πολύ. Θα θυμάστε ότι ασχοληθήκαμε ήδη ε, με το θέμα αυτό ε, ε, στη συνεδρίασή μας της 14 η Ιουνίου και ακολουθήσαμε την γρήγορη επίγουσα διαδικασία γιατί θεωρήσαμε ότι είναι σημαντικό θέμα. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Κομισιόν έτσι ώστε να μας δώσει κάποιες διευκρινήσεις για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρία Μάρκος. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να, να ευχαριστήσω ε, την Επιτροπή σας ε, που προσκάλεσε την ε, Κομισιόν σε αυτή τη συζήτηση. Αλλά τώρα θα συνεχίσω στα αγγλικά γιατί αυτή είναι η γλώσσα εργασίας και για να σεβαστώ τους διερμηνείς, λέει η ομιλήτρια. Κοιτάξτε, δεν είχαμε πάρα πολύ χρόνο γιατί ακολουθήσατε την επιτυχημένη διαδικασία. Εάν πραγματικά θέλετε ε, ε, να μελετήσει η Κομισιόν αυτήν την ε, αναφορά, τότε θα πρέπει να μας στείλετε και όλη, όλα τα σχετικά στοιχεία. Όσον αφορά ε, όσον αφορά τώρα το ίδιο το κλείσιμο της επιχείρησης, ε, βεβαίως ής ε, την, στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να κλείνουν αν πάρουν μια τέτοια απόφαση. Βεβαίως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα κοινωνικά ζητήματα τα οποία με, με την πάυση δραστηριοτήτων συνδέονται. Ωστόσο, η Κομισιόν καλεί όλους τους ε, ε, εμπλεκόμενους σε οποιαδήποτε διαδικασία αναδιάρθρωσης ε, να ακολουθούν τις καλύτερες δυνατές από κοινωνική και οικονομική άποψη δυνατότητες έτσι ώστε στην αναδιάρθρωση να δημιουργηθούν όσο γίνεται λιγότερα προβλήματα. Όλα αυτά αναφέρονται σε ανακοίνωση της Κομισιόν με ακριβώς το θέμα αυτό, δηλαδή την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων. Στην ουσία δηλαδή πρόκειται για κάποιες ε, πρακτικές ε, ε, οδηγίες που πρέπει να ακολουθούν οι επιχειρήσεις αλλά και οι εργαζόμενοι και οι δημόσιες τοπικές αρχές. Ε, το σημαντικότερο στοιχείο της ανακαυτής ε, είναι ε, η επιδίωξη της ευέλτης της δυνατής συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων σε τέτοιες διαδικασίες. Επίσης είναι σαφές ότι οπωσδήποτε θα πρέπει σύμφωνα και με, τον ευρωπαϊκό, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία να έχουν προηγηθεί από πλευρά των εργοδοτών διαβουλεύσεις ε, και συνεργασία ε, με τους ε, εργαζόμενους έτσι ώστε να είναι οι αποφάσεις συμβατές με το κεκτημένο. Επίσης ε, έχουμε και την οδηγία 9859 ε, η οποία αντιμετωπίζει το θέμα ε, και διευθετεί το θέμα των συλλογικών απολύσεων. Εκεί λοιπόν αναφέρεται ότι θα πρέπει οι αποφάσεις για συλλογικές απολύσεις να έχουν ληφθεί εν ευθέτω χρόνο, να έχουν, να έχουν μελετηθεί σωστά έτσι ώστε να μειώνεται στο μεγαλύτερο βαθμό ο αριθμός των ε, προσαπόληση εργαζομένων και επίσης ε, ότι θα πρέπει να προβλεφθούν συνοδευτικά κοινωνικά μέτρα. Κατά τα λοιπά, οι αρμόδιες εθνικές ε, αρχές, ε, ε, οι επιθεωρητές και τα δικαστήρια θα είναι υπεύθυνα για, την, για τον έλεγχο της σωστής εφαρμογής των, του κοινοτικού κεκτημένου και των νομοθετημάτων που έχουν ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία. Γνωρίζουμε ότι στην προκείμενη περίπτωση υπάρχει ε, μία ε, διαβούλευση η οποία ε, έχει ξεκινήσει ανάμεσα στη Χούντα, ανάμεσα δηλαδή στο Δημοτικό Συμβούλιο τους εργαζόμενους και, τους, την επιχείρηση και τους εργαζόμενους οπότε θα πρέπει να περιμένουμε και το αποτέλεσμα. Όσον αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιτροπή έχει δημιουργήσει τον ε, χάρτη της ε, κοινωνικά υπεύθυνη ε, στρατηγικής που βρίσκεται τώρα τελείως υπό αναθεώρηση. Ε, οπωσδήποτε υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές όσον αφορά το επιχειρήν και την, τις κοινωνικές συνθήκες που πρόκειται για κείμενο το οποίο ακολουθεί τις αρχές του ΩΣΑ. Ε, αλλά βεβαίως ε, ε, εδώ αναφερόμαστε σε δεσμεύσεις τις οποίες πρέπει να αναλάβουν όλες οι ενωσιακές επιχειρήσεις είτε δρούν στην την ενωσιακή επικράτεια είτε εκτός. Μιλάμε εδώ για δραστηριότητες οι οποίες ε, μπορούν να διευρύνουν ε, τον, την, τον επί, την κοινωνική επίπτωση ε, των αποφάσεων των επιχειρήσεων. Όσον αφορά τώρα τη, την πρόσβαση στα διαφορετικά ταμεία, σύμφωνα με την πρώτη έρευνα που έκανε η Κομισιόν, ε, τα τελευταία χρόνια η επιχείρηση αυτή δεν έχει λάβει, ε, δεν έχει λάβει ε, επιδοτήσεις από ευρωπαϊκά ταμεία, τουλάχιστον όχι από το 2014 και μέχρι σήμερα. Αλλά βεβαίως όταν θα έχουμε και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία στη διάθεσή μας θα προχωρήσουμε σε εντελεχέστερη μελέτη. Η Άγχελα πρώτα. Οι συνάδελφοι δηλαδή τώρα θα πάρουν το λόγο. Άγχελα. Ευχαριστώ, Σεσίλια. Εμείς υποστηρίξαμε αυτή την αναφορά ε, βάσει της ε, επίγουσας ε, διαδικασίας γιατί θεωρούμε γιατί θεωρούμε ότι το ζήτημα είναι σημαντικό. Ε, κοιτάξτε, ε, αυτό το εργοστάσιο και λόγω μεγέθους και λόγω ιστορίας είναι σημείο αναφοράς στην ε, περιφέρεια Καστιγιά ε, η Λέων και επομένως έχει συμβάλει σε πολλές θέσεις εργασίας άμεσης και έμεσης. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα της σταδιακής απορρίθμισης των τέτοιου είδους εργοστασίων και εγκαταστάσεων που αφορούν ε, τον ε, ε, γεωργικό, τροφιμικό, κτηνοτροφικό τομέα. πρέπει να ξέρουμε να μάθουμε εάν έχει πάρει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση η εταιρεία αυτή και πώς τη χρησιμοποίησε. Πρέπει να μελετήσουμε σε βάθος το θέμα αυτό. Και επίσης νομίζω ότι θα πρέπει όντως να μελετήσουμε σε βάθος το θέμα για να δούμε εάν υπάρχουν ε, ε, στοιχεία και συμπεριφορές ασύμβατες με την αρχή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Νομίζω ότι από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης θα πρέπει ε, να ξαναδούμε λίγο τα, την αποβιομηχάνηση και την πίεση την οποία δέχεται η εργατική τάξη σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα ε, να ε, αναφέρω ότι η ε, ΓΚΟΕ, η Ενωτική Αριστερά, Ευρωπαϊκή και Ισπανική, στηρίζει την, τους εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Εδώ βλέπουμε μια περίπτωση γνωστής συμπεριφοράς γιατί έχουμε μελετήσει εδώ στην Επιτροπή Αναφορών παρόμοιες περιπτώσεις και στο παρελθόν. Ε, δηλαδή ε, επιχειρηματίας ο οποίος σιγά σιγά ε, μεταφέρει τις δραστηριότητες από ένα εργοστάσιο σε ένα άλλο χωρίς να σκεφτεί καθόλου τις κοινωνικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει για τους εργαζόμενους αλλά και για την περιοχή μεταφορά λοιπόν της ε, ε, παραγωγής από το ένα εργοστάσιο στο άλλο με μόνο γνώμονα το κέρδος ε, και εδώ, ε, στην προκείμενη περίπτωση, το ίδιο συμβαίνει. Θα μείνουν χωρίς δουλειά τόσοι άνθρωποι ε, και εδώ μιλάμε για, μια, για ένα εργοστάσιο το οποίο δεν υπέφερε καθόλου οικονομικά, δεν είχε καθόλου οικονομικές απώλειες. Θα πρέπει να μελετήσουμε το θέμα σε σχέση με τις επιδοτήσεις από τα διορθωτικά ταμεία, να δούμε εάν χρησιμοποιήθηκαν οι πόλοι Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε να έχουν χρησιμοποιηθεί ευρωπαϊκά χρήματα από τα διορθωτικά ταμεία έτσι ώστε να υποβοηθηθεί το κλείσιμο μιας ε, ε, επιχείρησης ε, χωρίς ε, οικονομικό λόγο. Ε, θα πρέπει να τα δούμε λοιπόν, οπωσδήποτε δεν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτό το κλείσιμο και αυτή η διαδικασία γίνεται δυνατή λόγω των αποφάσεων των οποίων έχει πάρει η Ισπανική κυβέρνηση, λόγω των αποφάσεων που έχει πάρει το, Ευρωπαϊκό, συγγνώμη, το Ισπανικό Λαϊκό Κόμμα που δίνει την δυνατότητα να, να παίρνονται αυτές οι αποφάσεις από πλευράς ε, των επιχειρήσεων ε, και που δίνει τη δυνατότητα να μείνουν τόσοι άνθρωποι χωρίς δουλειά. Θα πρέπει κατά αυτή την έννοια να, να μεταφέρουμε το θέμα και στην κοινωνική υπηρεσία και, και, η Επιτροπή, και η Επιτροπή Απασχόλησης. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ δεν θέλω να γίνει πολιτική συζήτηση η εν μέρη πολιτική συζήτηση. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να σεβαστούμε ε, τον αναφέροντα και να μην μπούμε σε πολιτικές συζητήσεις, ούτε να βάλουμε πολιτικές ετικέτες, ούτε να δείχνουμε με το δάχτυλο κάποια πολιτικά κόμματα. Ε, The floor is yours. Και πρώτη φορά βλέπω τον κύριο Ριμέρα εδώ και του δίνω το λόγο. Χαίρομαι, χαίρομαι. Χαίρομαι που σε βλέπω και εδώ αγαπητή Σεσίλια. Βλεπόμαστε σε άλλες επιτροπές. Παρατήρηση εκτός μικροφώνου. Λοιπόν, τώρα θα αρχίσουμε, τώρα θα αρχίσει να μετράει ο χρόνος μου κυρία Πρόεδρε, γιατί εγώ πριν απάντησα στον κύριο Φερνάνδο Κάβρας. Όπως και υπόθηκε προηγουμένως, το, και σημαντικό, ε, το σημαντικό της σημερινής συζήτησης είναι η προστασία των εργαζομένων στο ίδιο το εργοστάσιο ε, ε, επεξεργασίας γάλακτος, αλλά και στους περίπου 100 κτηνοτρόφους, των οποίων η δραστηριότητα σχετίζεται άμεσα με αυτό το εργοστάσιο. Ε, σταματάει λοιπόν η δραστηριότητα και έχουν επιπτώσεις όλοι αυτοί οι άνθρωποι χωρίς όμως ε, καμία ε, αιτιολόγηση. Τα τελευταία χρόνια ο Όμιλος ε, Λακτάλης ε, έχει κάνει ε, πάρα πολλά στραβά βήματα. Πιστεύουμε δε ότι θα πρέπει να μελετηθούν ιδιαιτέρως όλες οι αποφάσεις του Ομίλου Λακτάλης και αν προκύψουν παρανομίες ή παραβάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κινηθεί άμεσα. Θα πρέπει επίσης να μελετηθεί η ενδεχόμενη ή η ενδεχομενη η εδω ε, αναφερόμενη κακή χρήση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ε, ε, η οποία ενδεχομένως βοήθησε να βελτιωθούν κάποια εργοστάσια προς ζημίαν του εν λόγω εργοστασίου. Εάν συνέβη κάτι τέτοιο το καταγγέλουμε ή το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι, ε, ε, ε, η Δημοτική Αρχή της περιοχής αλλά και η Ένωση για την διατήρηση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή από κοινού αντιμετωπίζουν το θέμα σημαίνει ότι θα πρέπει να το δούμε και εμείς από κοντά. Δεν είναι δυνατόν να δικαιολογηθεί με κάθε τρόπο η μ ε, μαζική απόλυση τόσων εργαζομένων και οπωσδήποτε δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτήν την συνολική, τη συλλογική απόλυση ε, που ενδεχομένως έχει προκύψει μόνο διότι η επιχείρηση αποφάσισε ε, απλά να μεταφέρει τις δραστηριότητες αλλού. Στην Καστίγια Λεών όπως είπα και προηγουμένως, όλες οι αρχές και όλες οι πολιτικές δυνάμεις ενώνονται έτσι ώστε να υποστηρίξουν τους εργαζόμενους σε αυτό το εργοστάσιο. Εργοστάσιο το οποίο θα πρέπει να παραμείνει, να συνεχίσει τις δραστηριότητες ε, ε, του. Ε, είπα και προηγουμένως ότι θα πρέπει να μελετηθεί η κατάσταση του ομίλου Λακτάλης έτσι ώστε να ληφθούν οι αποφάσεις αυτές οι οποίες θα επιτρέψουν στους εργαζόμενους να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Στρέφαμε προς την Κομισιόν. Ε, Βεβαίως ε, εκτιμώ θετικά την προσπάθειά σας να δώσετε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ε, μια δομημένη απάντηση. Αλλά το είπατε κι εσείς αγαπητή κυρία, δεν έχετε τα απαραίτητα στοιχεία, δεν έχετε όλα τα στοιχεία αυτά που θα σας δώσουν την δυνατότητα να απαντήσετε ε, απολύτως αιτιολογημένα. Θα πρέπει λοιπόν και οι πολιτικές ομάδες και οι εργαζόμενοι και οι το Δημοτικό Συμβούλιο να στείλουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Απ' την άλλη πλευρά, πρέπει να σας πω το εξής. Αναφερθήκατε στην εντελική κοινωνική ευθύνη. Ε, είναι, υπάρχει πληθώρα δηλώσεων ε, από τις κοινωτικές αρχές ε, και πληθώρα ε, και πληθώρα δηλώσεων υπέρ της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και υπέρ των κοινωνικών δικαιωμάτων των ε, εργαζομένων. Εσείς αγαπητή κυρία αναφερθήκατε στην ε, ελεύθερη διακίνηση και στην ελευθερία εγκατάστασης. Ωραία, έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά, αλλά δεν υπάρχει στην, στις αρχές και στα κείμενα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα καμία παράγραφος η οποία ε, να ε, λέει ε, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν με άλλο τρόπο τα ευνοσιακά ευρωπαϊκά κονδύλια. Επίσης αναφερθήκατε στην οδηγία 9859 αλλά καταλαβαίνετε ότι στην προκείμενη περίπτωση δεν ισχύει ε, δεν ισχύουν ε, τα, τα κείμενα αυτά γιατί εδώ έχουμε προσχεδιασμένη και αδικαιολόγητη ε, απομάκρυνση και απόλυση των εργαζομένων. Ε, ολοκληρώνω κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι θα πρέπει να σταλθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλα αυτά τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία θα της δώσουν τη δυνατότητα να έχει μια πιο ολοκληρωμένη άποψη και επομένως να τροποποιήσει την αντιμετώπιση της ε, όσον αφορά το θέμα αυτό. Ευχαριστώ, Όταν μιλάς ε, ισπανικά, ε, πραγματικά νιώθω ότι αποτελεί έλλειψη από τη δική μου ε, πλευρά το ότι δεν μπορώ να καταλάβω ισπανικά αλλά και η διερμηνία είναι πάρα πολύ καλή οπότε τους ευχαριστώ και τους διερμηνείς ε, για αυτήν την τόσο αναλυτική παρουσίαση. Ο λόγος όμως τώρα στην κυρία Πιτέρα. Ευχαριστώ. Ε, νομίζω πως αυτό το ζήτημα ακόμα δεν μπορούμε να το εξετάσουμε οριστικά γιατί ακούω ε, τα όσα μας λένε εκπρόσωποι εδώ ε, από την πλευρά του αναφέροντος ακούω τα όσα μας λέει η Επιτροπή για το ότι αυτή η επιχείρηση από το 2014 δεν έχει αξιοποιήσει ευρωπαϊκά κονδύλια και θέλει να το εξετάσει περαιτέρω οπότε ενδεχομένως θα πρέπει να δούμε αυτή την πτυχή και θα ήθελα επίση να μάθω ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να μετακατασταθεί εν λόγω μονάδα. Γιατί βέβαια μπορούν να υπάρχουν μια σειρά από διαφορετικοί λόγοι. Μπορεί δηλαδή να, η μετακατάσταση να συνεχίζεται με λόγους μεγιστοποίησης των κερδών, αλλά θα μπορούσε να υπάρχει για παράδειγμα κίνδυνο επτόχευσης ε, για, το για τη συγκεκριμένη μονάδα ή για ολόκληρη την επιχείρηση, πράγμα βέβαια το οποίο θα οδηγούσε στην ε, αναγκαστικά σε ακόμα πιο μεγάλη μείωση των θέσεων εργασία. Οπότε επειδή δεν γνωρίζουμε τους λόγους θα πρέπει να το δούμε περαιτέρω. Ε, Ευχαριστώ. Σταρές τώρα. σα ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα να καλωσορίσω ε, την Μιλάγρος ε, Μάρκος ε, και την ομάδα της. Όλες οι πολιτικές ομάδες της ε, Καστίγιας ε, Λεών εκπροσωπούνται στην, ε, στο Δημοτικό Συμβούλιο του οποίου εκπρόσωπος είναι η κυρία Μιλάνδρος. Υπάρχουν τρία θέματα τα οποία αντιμετωπίστηκαν εδώ και τα οποία είναι σημαντικά για μένα. Πρώτα απ' όλα η παραβίαση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, 85 εργαζόμενοι καθώς επίσης και οι κτηνοτρόφοι και όλοι οι, άμεσα, οι έμεσα εμπλεκόμενοι χάνουν την δουλειά τους τρόπο προσχεδιασμένο και αδικαιολόγητο ε, λόγω αυτής ε, της ε, μετεγκατάστασης. Είδαμε ότι σε αυτό το εργοστάσιο του Βαγιαδολίδη η παραγωγή μειωνόταν με προσχεδιασμένο τρόπο. Υπάρχει όμως και ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα. Είναι αυτό των διορθωτικών ταμείων. Τα, τα ταμιά ταμεία και τα ταμεία συνοχής είναι τα ταμεία τα οποία δημιουργήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να συμβάλλουν στην συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοχή η οποία συνδέεται με τα κοινωνικά, με την ελληνική αλλά και με την ανάπτυξη εδώ συμβαίνουν ακριβώς τα αντίθετα. Βλέπουμε μία προσχεδιασμένη ε, μετεγκατάσταση που αντιτίθεται ε, εις ε, τους στόχους της ανάπτυξης, της προώθησης, της προόδου το, μέσω των διευθυντικών ταμείων. Άρα αντιτίθεται αυτή η διαδικασία στο μέλλον της συνοχής. Μέσω λοιπόν των χρημάτων των ταμείων εδώ βλέπουμε ε, ε, ε, γίνονται ε, πράγματα τα οποία σαφέστατα έρχονται σε αντίθεση με τις αρχές που διέπουν υποτίθεται τα μία αυτά. Και τέλος το θέμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Αυτό είναι ένα άλλο από τα κεντρικά, τα εμβληματικά στοιχεία ε, και του Κοινοβουλίου ε, εντός της ε, ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο που είναι αυτή η εταιρική κοινωνική ευθύνη. Χαιρόμαστε που έχουμε εδώ την εκπρόσωπο του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία ταυτόχρονα εκπροσωπεί επομένω όλε τι πολιτικέ δυνάμει αλλά εκπροσωπεί ε, και αυτήν την ε, ε, υπηρεσία για την παραμονή τη επιχειρηματικότητα στην επικράτεια τη Καστίγια Ελαιών. Και επομένω δεν υπάρχει κανένα λόγο να πούμε ότι δεν είμαστε αρμόδιοι εδώ. Βρισκόμαστε κατάφορα απέναντι σε ένα θέμα το οποίο είναι αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Οι εργαζόμενοι, οι, κοινωνία, το, οι, οι πολίτες θα πρέπει να κατανοήσουν ότι η Ευρώπη είναι εκεί για να τους βοηθήσει και ότι ε, μπορεί να βοηθήσει την οικονομία, μπορεί να βοηθήσει την κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σουσακάρη Κάμπρας. Και κλείνει εδώ ο κατάλογος ομιλητών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα ισπανικά. Γιατί ξέρετε έχουμε πολύ καλούς διερμηνείς, λέει που ε, καλύπτουν αυτό το γλωσσικό χάσμα μεταξύ μας. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω εξ των, ε, ε Πρασίνων. Ε, η αναφέρουσα αναφέρθηκε σε τρία στοιχεία τα οποία προσυπογράφω. Αλλά νομίζω ότι εδώ έχουμε ένα απολύτως θεμελιώδες ζήτημα. Όλοι δεχόμαστε τον καπιταλισμό. Ωραία και ο καπιταλισμός είναι σκληρός και κάθε μέρα γίνεται σκληρότερος. Το δείχνει και η Κομισιόν με τα, σχόλια που έκανε, γιατί μας είπε εταιρική κοινωνική ευθύνη, αλλά ναι μεν αλλά και διάφορα, διάφορες ρητορικές ε, περικοκλάδες και το αποτέλεσμα ποιο είναι, ότι την πατάει ο εργαζόμενος. Ε, με τον Αγκουστίν, με την Άγχελα, με τη Μαρίνα, με όλους τους συναδέλφους μου, ε, και με όσα αυτά που ε, μόλις είπαν ε, οδηγούμαστε στο ότι θα πρέπει κυρίως να ασχοληθούμε με το δεύτερο σημείο που αναφέρατε αγαπητή κυρία που είναι το θέμα της εσφαλμένης χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων γιατί διαφορετικά θα μας ξεφύγουν οι υπεύθυνοι εάν αρχίζουμε να μιλάμε για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και για τα άλλα κοινωνικά. Κοιτάξτε, όλα τα υπόλοιπα, ε, ηθικά και πολιτικά, όλα τα στοιχεία που αναφέρατε είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ε, αυτά δεν τα καταλαβαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι καπιταλιστές όλοι. Ε, και το λέω με συμπάθεια. Όχι συμπάθεια προς τον καπιταλισμό, συμπάθεια προς τον εκπρόσωπο, την χαριεστάτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό το δεύτερο σημείο το οποίο αναφέρατε. Να δούμε χρησιμοποιήθηκαν σωστά ή εσφαλμένα τα υπόρρητα των διορθωτικών ταμείων. Ευχαριστώ. Όλο ένα και πιο εμφάνταστη και δημιουργική γινόμαστε στην Επιτροπή. Να δώσουμε τώρα το λόγο στην αναφέρουσα για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ όλους ε, για τις παρεμβάσεις σας. Ε, πρώτα απ' όλα, πιστεύω ότι η προσχεδιασμένη μετεγκατάσταση ε, οπωσδήποτε ε, έχει βασιστεί ή εν πάση περιπτώσει έχει οδηγήσει σε προσχεδιασμένη συλλογική απόλυση. νομίζω ότι και η έκθεση αυτής της, της του οργανισμού Ανκλάχ Πρεσαριάλεο την οποία εκπροσωπώ ε, αναφέρει ότι είναι απολύτως ανταγωνιστική αυτή ε, η, αυτό το εργοστάσιο του συγκεκριμένου ομίλου ε, και επομένως δεν δικαιολογείται αυτή η μετεγκατάσταση η ανταγωνιστικότητα και η αποτελεσματικότητα αυτού του εργοστασίου του Βαγιαδολίθ δεν τίθενται υπό αμφισβήτηση αντιθέτως επειδή είναι από τις πιο παλιές εγκαταστάσεις ε, σίγουρα το μισθολογικό κόστος είναι μεγαλύτερο. Όντω το, το σημείο το δεύτερο αυτό των ε, ε, ταμείων ε, πρέπει να μελετηθεί γιατί εμείς θα πρέπει να μελετήσουμε το κατά πόσον στο παρελθόν αλλά τώρα αλλά και στο μέλλον γιατί και η πρόληψη είναι πολύ σημαντική πρέπει να προλαμβάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς γνωρίζουμε, έχουμε λάβει γνώση του γεγονότος ότι έχει λάβει ο όμιλος αυτός ε, ε, επιδοτήσεις ε, και κονδύλια από τα διορθωτικά ταμεία. Θα πρέπει να μελετηθεί λοιπόν πώς χρησιμοποιήθηκαν τα, τα, τα, χρήματα αυτά. Γιατί εάν χρησιμοποιήθηκαν πόροι από τα διορθωτικά ταμεία έτσι ώστε πόροι οι οποίοι θεωρητικώς βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να αναπτύξουν την ύπεθρο, έτσι ώστε να βελτιώσουν τη συνοχή, να βελτιώσουν την διάσταση μεταξύ διαφορετικών περιοχών. Εάν λοιπόν χρήματα από αυτά τα διορθωτικά ταμεία έχουν χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε ε, να, χρηματοδοτηθούν άλλα ε, εργοστάσια και να οδηγήσουν στη μεταγκατάσταση και το κλείσιμο αυτών των, ε, του εργοστασίου στο βαγιαδολίθε τότε αυτό θα πρέπει να μελετηθεί ενδελεχώς. Όσον αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη, θεωρούμε ότι και εδώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. από πλευράς του ομίλου Λακτάλης δεν είχαμε καμία κοινωνική μέρημνα, δεν είχαμε καμία ευαισθησία κοινωνική ή εργασιακή ε, αυτή τη στιγμή απολύονται οι εργαζόμενοι και ακόμα περισσότερο απαγορεύεται η πώληση αυτού του εργοστασίου ε, σε κάποιον τρίτο ενδιαφερόμενο ε, με μόνο σκεπτικό την μείωση του ανταγωνισμού από πλευράς του ομίλου λακτάλισε. Ε, θα πρέπει τουλάχιστον να επιτραπεί η πώληση σε κάποιο ενδεχόμενο ενδιαφερόμενο ο οποίος ενδεχομένως θα αναλάβει ε, και την, ε, ορισμένους από τους απολυμμένους εργαζομένους. Γι' αυτό λοιπόν φτάσαμε εμείς εδώ γιατί καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο της δικής μας περιοχής μπορεί και σε άλλες περιοχές σε άλλοι εργαζόμενοι να υποφέρουν από παρόμοιες καταστάσεις. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε ε, και τώρα αλλά και στο μέλλον να αποφευθούν τέτοιου είδους καταστάσεις ε, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε εσφαλμένη και εγκληματική από κοινωνική και οικονομική απόψεως και από απόψεως συνοχής ε, χρήσης των πόρων των διαχρονικών ταμείων. Νομίζω ότι εδώ ε, χρειαζόμαστε μία ε, ελπίδα να δώσουμε σε αυτούς τους 85 άμεσα εργαζόμενους και τους 100 έμεσα εμπλεκόμενους εκτινοτρόφους και τις οικογένειές τους. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Σας διαβεβαιώνω ότι Σχεδόν ποτέ δεν υπάρχει απόλυτη ομοφωνία στην Επιτροπή από όλε τι πολιτικέ ομάδε. Και όμω σήμερα συνέβη. Δεν συμβαίνει συχνά, να ξέρετε. Μπορείτε λοιπόν να επιστρέψετε στην περιφέρειά σα και να μεταφέρετε το μήνυμα στους εργαζομένους ότι η Επιτροπή Αναφορών ομοφόνος σας έχει στηρίξει και έχει στηρίξει την υπόθεση των εργαζομένων. Θα ήθελα όμως ε, να επισημάνω την εξή διέξοδο. Προτείνω λοιπόν εσεί όσο αναφέρουσα εξ ονόματο των εργαζομένων να στείλετε επιπλέον πληροφορίες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς την Γραμματεία της Επιτροπής μας εδώ προκειμένου να διερευνήσουμε περαιτέρω κατά πόσο τα δραστικά ταμεία την χάνουν κατάχρηση εδώ. Είναι η μοναδική νομική οδός που μπορούμε να ακολουθήσουμε για να δούμε αν, υπάρχουν, ε, αν υπάρχει παραβίαση των ευρωπαϊκών κανόνων για την χρήση των διεθνωτικών ταμείων και των περιφερειακών ταμείων. Και αν ε, αντιβαίνουμε έτσι στις αρχές της ε, συνοχής και αλληλεγγύης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι μια πρόταση λοιπόν και μετά μπορούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ρωτήσουμε, να απαντήσει μάλλον εκείνη αν ε, ισχύει κάτι τέτοιο ή όχι. Στο Κοινοβούλιο η κοινωνική εταιρική ευθύνη, όμως ομως δυστυχώ, δεν είναι υποχρεωτική, είναι εθελοντική. Προαιρετικά λοιπόν οι επιχειρήσεις επιλέγουν να εφαρμόσουν ένα σύνολο κανόνων, αλλά δεν είναι δεσμευτικό όλο αυτό, δεν μπορούμε να νομοθετήσουμε, μπορούμε μόνο να το προωθήσουμε ως ε, καθεστώς. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλές βέβαια στο Κοινοβούλιο και το βλέπετε αυτό σε πολλές επιτροπές. Εδώ γίνεται λόγος για μια ιδιωτική επιχείρηση και αυτό είναι απόφαση της διοίκησης. Επομένως ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσημη αρμοδιότητα να παρακάμψει τις αποφάσεις ε, τη διοίκηση μια επιχείρηση. Όμως μπορούμε και πάλι να του πούμε ότι δεν εγκρίνουμε αυτή του τη στάση. Σας καλούμε λοιπόν να επανέλθετε με περισσότερες πληροφορίε, βεβαίω θα διατηρήσουμε ανοιχτή την αναφορά. Υπάρχει συνεχής διάλογος και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε κατά πόσο γίνεται κατάχρηση των ε, Ευρωπαϊκών Ταμείων ή όχι και μετά μπορούμε να έρθουμε απευθείας σε επαφή με τη διοίκηση της επιχείρησης. Όμως, είναι πραγματικά μια ιστορική στιγμή στην Επιτροπή Αναφορών, όπως προανέφερα, ότι για πρώτη φορά είμαστε ενωμένοι και από κοινού όλοι στηρίζουμε την υπόθεσή σας. Σας ευχαριστώ που ήρθατε μέχρι εδώ. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο μέλλον για μια περιφέρεια της Ευρώπης που από ό,τι ξέρω είναι πανέμορφη. Σας ευχαριστώ. Ας περάσουμε τώρα στην 259 αναφορά, επίσης ισπανική, από την Ασοσιασιόν Σαλβάρ Λατεχίτα στην Τενερίφη. Τι ωραία. Βίβα Ισπάνια. Πάνω πήγα να πω να δώσουμε το λόγο στην αναφέρουσα για πέντε λεπτά. Η πλατφόρμα Σαλβάρ Λατεχίδα ε, δημιουργήθηκε με στόχο την διάσωση της εμβληματικής ε, ε, παραλίας Λατεχίδα καθώς επίσης και του ειδικού εθνικού δρυμού του, της Μοντάνια Ρόχα και είναι ένα από τα πιο όμορφα σημεία και τις πιο όμορφες τοποθεσίες της Τενερίφης στα Κανάρια νησιά και που κινδυνεύει να αντιμετωπίσει μεγάλη μεγάλο λόγω της οικοδόμησης μιας μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας. <clears throat> Ε, η Μοντάνια Ρόχα ονομάστηκε Εθνικός Δρυμός από το 1987 βάσει του νόμου 12 του 1987 και ε, άρχισε να συμμετάσχει στο δίκτυο των Καναρίων των προστατευμένων ε, φυσικών τοποθεσιών. Ήδη από το δε ε, έχει ταξινομηθεί ως, ειδική, ε, ως ειδικός ε, εθνικός βιότοπος. Ε, πρέπει να πούμε ότι ε, αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα κυριότερα στοιχεία ε, τουριστικού ενδιαφέροντος που το αντιμετωπίζουν με εξαιρετικό ενδιαφέρον οι τουρίστες ήδη της δεκαετίας του 70 και του 80. Η παραλία της Λατεχίτα που ανέφερα προηγουμένως καθώς επίσης και ο ειδικό δρυμός, ο προστατευμένος δρυμός της Μοντάνια Ρόχα έχουν μέχρι τώρα διασωθεί. Ε, έχουν δε καθοριστεί ως ειδικέ ε, ε, περιοχές προστασίας. Πρόκειται κυρίως για ειδική ζώνη συντήρησης μέσα στην ρεχιόν Μακαρονέσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν πουλιά όπως το τσορλιτέχο πατινέγρο που ε, κινδυνεύουν να εξαλειφθούν. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και άλλα ε, τα οποία έχουν ήδη εξαφανιστεί. Πέρα από αυτό όμως θεωρούμε ότι ο βαθμός ε, συντήρησης είναι πάρα πολύ ελλειπής Πρέπει εδώ να πούμε επίσης ε, ότι ε, στο Σαβαδάλες Δελσούρντε Τενερίφε είναι μια ε, παραλία, μια τοποθεσία θαλάσσια η οποία επίσης είναι καταγεγραμμένη ως ειδική ζώνη συντήρησης. Αυτό λοιπόν το φυσικό ε, σύμπλεγμα το οποίο δημιουργείται από την παραλία της Τεχίτα και από το κόκκινο φουνό αυτήν την Μοντάνια Ρόχα, ε, ε, είναι ιδιαίτερα προσφυλής σε όλους τους κατοίκους του, της νότιας Τενερίφης αλλά και σε όλους τους κατοίκους του νησιού καθώς επίσης και στους τουρίστες. Σε αυτό το ιδιαίτερα οικολογικό και όμορφο περιβάλλον προβλέπεται η κατασκευή ενός ξενοδοχείου σε 26.000 τετραγωνικά μέτρα σε τρία επίπεδα τα οποία θα, το οποίο θα έχει 312, 312 ε, δωμάτια και χωρητικότητα 800 κλινών. Προβλέπεται δε η οικοδόμηση δίπλα ακριβώς στην προστατευμένη περιοχή ε, δεν είναι δυνατόν να επιτραπεί επομένως κάτι τέτοιο. Ε, πρέπει εδώ να προσθέσουμε και το μεγάλο πρόβλημα ε, της αποχέτευσης που ήδη είναι ιδιαίτερο βαρύ στην περιοχή της Γραναδίγια Ντεαμπόνα και όπου οπωσδήποτε θα επιβαρυνθεί. Κατά αυτή την έννοια θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι η οδηγία Habitat 9243 της ΕΟ και το άρθρο 6 αναφέρει ρητά ότι οποιοδήποτε σχέδιο ή πρόγραμμα το οποίο ε, μπορεί να έχει επίπτωση στο ε, δίκτυο Natura 2000 θα πρέπει οπωσδήποτε να υπόκειται σε εκ των προτέρων ε, αξιολόγηση. Ε, ε, κατά την άποψή μας δεν είναι δυνατόν να επιτραπεί μια κατασκευή, μια δόμηση με τέτοια χαρακτηριστικά ε, σε ένα φυσικό περιβάλλον σαν αυτό που αναφέραμε προηγουμένως, δηλαδή αυτό της Μοντάνια Ρόχα από πλευράς Χερσαίας και από το Σεβαδάλες Δελσούρντε Τενερίφε από πλευράς Θαλάσσιας. Θέλουμε επίσης να αναφέρουμε ότι αυτή η κατάσταση δεν συνάδει με τα άρθρα 3 και 4 της Οδηγίας 2000 2009 ε, ε, Παύλα 147 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30 Νοεμβρίου του 2009 ε, που αναφέρεται κυρίως στα ενδυμικά πτηνά. Ε, ε, όλες οι οδηγίες ε, οι οποίες αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθηθεί η πρόταση της πλατφόρμας Αλβάρλα Τεχίδα. Η πλατφόρμα λαμβάνοντας υπόψη τις εν λόγω οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη επίσης τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει η περιοχή οδηγείται στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει έστω μια ενδιάμεση ζώνη επομένως κάποια μεταβατικά ενδιάμεσα ε, τμήματα τα οποία θα οδηγήσουν ε, σε ε, καλύτερη προστασία των περιοχών αυτών. Θέλουμε να σας πούμε επίσης ότι η πλατφόρμα έχει ήδη 100.000 υπογραφές οι οποίες οδηγούν, οι οποίες συμφωνούν με την στήριξη του δικού μας προγράμματος. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ανταποκριθεί στα αιτήματά σας και επίσης ε, το θέσαμε ως επίγον το ζήτημα μέσω απόφασης τον Ιούνιο. Και ξέρετε, δεν συμβαίνει πολύ συχνά αυτό. Θεωρήσαμε παραδεκτή την αναφορά και κινήσαμε την ταχύτερη δυνατή διαδικασία για να την εξετάσουμε. Στέφομαι τώρα στην Επιτροπή για να μας δώσει τυχόν νέες πληροφορίες για την υπόθεση και μια ενημέρωση για την σημερινή κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Όπως ε, είπαν ε, και οι αναφέρουσες έχουμε εδώ ε, ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα το οποίο θα ε, χτιστεί δίπλα σε δύο ε, τοποθεσίες οι οποίες συνδέονται, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο δίκτυο της Natura 2000 το, την Μοντάνια Ρόχα και τα Σαβαδάλες de Tenerife είναι γεγονός ότι οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους δεν ε, έδωσαν την απαραίτητη άδεια ε, σε αυτό το ε, σχέδιο και ε, ε, στην προκείμενη περίπτωση θα πρέπει να εφαρμοστεί το άρθρο 6 της οδηγίας Habitat ε, σύμφωνα με την οποία ρητά αναφέρεται ότι οποιοδήποτε σχέδιο μπορεί να έχει επίπτωση σε κάποια τοποθεσία του δικτύου που εμπίπτει στο Natura 2000 θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο πρώτερης αδειοδότησης και η αδειοδότηση μπορεί να δοθεί μονάχα εάν η εκ προτέρων αξιολόγηση ε, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν θα υπάρξει καμία ζημία προς ε, την ε, προστατευόμενη περιοχή. Εδώ δεν έχουμε αδειοδότηση και επίσης πριν από την ε, ε, ενδεχόμενη αδειοδότηση είναι βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα έχει ελέγξει ε, η Ισπανική κυβέρνηση αρμοδίως και ενδελεχώς την, το εν λόγω οικοδομικό σχέδιο έτσι ώστε να μην δώσει την αδειοδότηση σε περίπτωση κατά την οποία παραβιάζονται οποιαδήποτε αρχές σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Οπωσδήποτε δεν πρέπει να λησμονούμε ότι τα κράτη-μέλη είναι ε, οι κύριοι και πρώτοι υπεύθυνοι για την εφαρμογή της ε, νομοθεσίας έτσι όπως έχει μεταφερθεί και ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία και επομένως ε, ε, οι Ισπανικές αρχές θα είναι υπεύθυνε για την ε, τελική απόφαση για αυτού του σχεδίου. Όσον αφορά την δημιουργία ενδιάμεσων ζωνών, buffer zones, σε σχέση με τις προστατευόμενες περιοχές, δεν προβλέπεται αυτού του είδου η ζώνη στα πλαίσια του Natura 2000. Ωστόσο, το άρθρο 6 της οδηγίας Habitat ε, εφαρμόζονται ε, σε οποιοδήποτε σχέδιο ε, μπορεί να έχει οποιαδήποτε περιβαλλοντική επίπτωση σε περιοχές προστατευόμενες από το δίκτυο και από τη στιγμή που ε, ε, διαπιστώνουμε ότι κάποιο ε, σχέδιο οικοδομικό ή άλλο μπορεί να έχει ζημιογόνο επίπτωση σε προστατευόμενες περιοχές λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα. Τώρα, η Κομισιόν διευκρινίζει ότι η περιοχή ε, γύρω από την ε, παραλία της ε, Τεχίδα δεν έχουν ενσωματωθεί εις το πρόγραμμα Natura 2000. Σε αυτήν την περίπτωση τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία αποφασίζουν ποια είναι τα, ποιες είναι οι τοποθεσίες που προτείνονται για να ενσωματωθούν στο ε, δίκτυο προστασίας Natura 2000. Ε, ε, φτάνουν στην τελική τους απόφαση τα κράτη-μέλη στην επικουρούμενα από επιτροπές εμπειρογνωμόνων κτλ. και υποβάλλονται οι τοποθεσίες ή οι περιοχές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία λαμβάνει την τελική απόφαση λαμβάνοντας κυρίως υπόψη της ε, μια γενικότερη λογική και μια συνεκτική αντιμετώπιση ε, των ε, προστατευόμενων περιοχών σε τέτοια περίπτωση η Κομισιόν προχωράει σε τακτική αξιολόγηση έτσι ώστε να λάβει υπόψη τις προτάσεις οι οποίες αφορούν τα ενδιαιτήματα και τους βιοτόπους και την προστασία των ειδών και λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της για την ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κατανοεί ε, γιατί θα πρέπει ε, η παραλία της Λατεχίτα να ενσωματωθεί ε, σε μια ενδεχομένως διευρυμένη περιοχή προστασίας σύμφωνα με το Natura 2000. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχουν συνάδελφοι. Ο Χουάν Φερνάντο πρώτος. αν δεν σας πειράζει, ο κύριος Αφρόντε πρέπει να φύγει σε λίγο. Να του δώσουμε λοιπόν πρώτα το λόγο. Και μετά θα συνεχίσουμε με τον κατάλογο μιλητών. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δώσατε τον λόγο πρώτος γιατί πραγματικά πρέπει να φύγω. Ε, εγώ θα ήθελα να υποστηρίξω τα αιτήματα της πλατφόρμας Αρβάρα Τεχίτα γιατί εδώ καταστρέφουμε το περιβάλλον και την φυσική δομή του περιβάλλοντος ε, λόγω ε, της υποστήριξης ενός συγκεκριμένου ε, αναπτυξιακού ξενοδοχειακού μοντέλου. E Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η περιοχή αυτή, είναι ιδιαίτερου περιβαλλοντικού, ε, ε, περιβαλλοντικής σημασίας και ιδιαίτερου φυσικού κάλους και επομένως θα πρέπει ε, να σταματήσουν τέτοιου είδους δραστηριότητες. Θα πρέπει οπωσδήποτε και η παραλία της Λατεχίτα καθώς επίσης και οι παρόμοιες περιοχές θα πρέπει να ελέγχονται ενδελεχώς πριν δοθούν άδειες οικοδόμησης. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε ε, η εκτίμηση του περιβαλλοντικού αντικτύπου να γίνεται σωστά ε, με τις απαραίτητες προϋποθέσεις έτσι ώστε να μην παραβιάζεται με κανέναν τρόπο η οδηγία Natura 2000. Επίσης οι Ισπανικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν την πλήρη συμμετοχή του κοινού που θα πρέπει να έχει γνώση και γνώμη όσον αφορά τις σχετικές αποφάσεις. Επίση, οι τοπικέ αρχέ θα πρέπει να καλύψουν όλε τι ε, άλλε προβλεπόμενε ε, προποθέσει, οι οποίε ε, από την οδηγία προβλέπονται και κυρίως τα όσα ρητά αναφέρονται στο άρθρο 6 του εν λόγω νομοθετικού κειμένου. Ε, και που μπορεί να μην περιλαμβάνουν απαραίτητα περιοχές ε, που άμεσα ενέχονται στην ε, Natura 2000 αλλά μπορεί λόγω της γυτνίασης να έχουν συγκεκριμένες επιπτώσεις. Τέλος θα θέλαμε να αναφέρουμε τον κύριο, την, την μεγάλη σχέση που έχουν και οι, οι οδηγίες οι οποίες αφορούν την προστασία των πτηνών και την προστασία των ενδιατημάτων τους και θα πρέπει οπωσδήποτε οπωσδήποτε να προστατέψουμε τα οποιαδήποτε στοιχεία σχετίζονται με το Νατήρια 2000. Χουάν Φερνάντο, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω κι εγώ ισπανικά. In the routine here, Spanish case. Primero, quiero agradecer, por supuesto, la... Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την uh, εκπρόσωπο της uh, πλατφόρμας Αλβάρλα Τεχίτα που βρίσκεται εδώ μεταξύ μας. Μακάρι αυτές οι περιοχές να ήταν καλύτερα ε, γνωστές και να ήταν και η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καλύτερα γνωστή παντού. Ε, η δυνατότητα που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τίνει ευήκονους σε αναφορές, σε ε, θέματα τα οποία προκύπτουν άμεσα από την από τους πολίτες, από την κοινωνία των πολιτών που κινητοποιείται για θέματα τα οποία έχουν και ευρωπαϊκή διάσταση και που αφορούν ε, τον δημόσιο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή εδώ η περίπτωση. Και επομένως, κατά αυτή την έννοια, οποιαδήποτε δράση σε ε, εθνική επικράτεια μπορεί ε, να ε, αποτελεί παραβίαση κοινοτικής νομοθεσίας όπως εδώ της οδηγίας για το, το Natura 2000 είναι ευρωπαϊκό ζήτημα. Εγώ είμαι Ισπανός πολίτης, είμαι μέλος του, της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκπροσωπώντας την Ισπανία αλλά εγώ ε, είμαι επίσης γόνος των Καναρίων νήσων, ζω εκεί και εκπροσωπώ ε, την περιοχή και επομένως πρέπει να σας πω ότι σε όλη την πολιτική μου ε, ζωή απέδωσα πάρα πολύ μεγάλη σημασία εις ε, την ε, καταπολέμηση της άνερχης δόμησης και των χωροταξικών παραβιάσεων που δημιούργησαν πάρα, προκάλεσαν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα στο νησί. Ο τουρισμός που βεβαίως αποτελεί την ραχοκοκαλιά της οικονομίας των στα Κανάρια νησιά, ε, ο τουρισμός, λέω, δεν θα πρέπει να αποβαίνει σε ζημία της προστασίας του περιβάλλοντος στα Κανάρια. Ε, γιατί το θέμα της προστασίας του ε, περιβάλλοντος είναι πάρα πολύ σημαντική. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι λόγω και της αυτόνομης κυβέρνησης έχει δοθεί ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην, σημασία, προστασία του περιβάλλοντος. Επομένως, η οικοδόμηση ενός τεράστιου ξενοδοχείου ε, ε, στην, ε, στα Κανάρια μπορεί να μην αλλάξει τρομερά τη χωροταξία. Αλλά εγώ διάβασα και μελέτησα προσεκτικά. Φαίνεται ότι μέχρι τώρα τα στοιχεία είναι θετικά όσον αφορά την περιβαλλοντική επίπτωση. Δηλαδή υπάρχουν θετικές εκθέσεις από από το Δημοτικό Συμβούλιο, από το Συμβούλιο της ε, τοπικής κυβέρνησης των Καναρίων, το τμήμα δηλαδή το οποίο ασχολείται ακριβώς ε, με την, ε, με την νομοθεσία της Ισπανίας όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την ιδιαίτερα αυστηρή ισπανική νομοθεσία, τη λεγόμενη Λέιντε Κώστας, η οποία διέπει την δόμηση στις, στην Αιγιαλίτιδα ζώνη. Πρέπει να σας πω ότι είναι ιδιαίτερα αυστηρός νόμος, απαγορεύει οποιαδήποτε οποιαδήποτε και προλαμβάνει οποιαδήποτε δόμηση ε, στην Αγιαλίτιδα ζώνη ή οποιαδήποτε δόμηση η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα στο θαλάσσιο περιβάλλον και εδώ βλέπουμε ότι καλύπτονται οι προϋποθέσεις ε, και της Λέιντε Κώστας. Ε, έχει λοιπόν την τελική, ε, το τελικό πράσινο φως από την υπηρεσία ε, της, των παραλιών και των αγελίδων, ζωνών. Βλέπουμε επίσης σύμφωνα με, το πράσινο φως το οποίο έχει δοθεί και από την τοπική κυβέρνηση και από το Δημοτικό Συμβούλιο ότι με κανένα τρόπο δεν έχει επίπτωση η οικοδόμηση του συγκεκριμένου ξενοδοχείου στη Μοντάνια Ρόχα, ούτε ε, στις ε, περιοχές ε, της Ρεζέρβα Naturale Special de Montaña ρόχα, ούτε και σε την περιοχή της, του δικτύου των Καναρίων σε σχέση με, την, με τα προστατευμένα φυσικά περιβάλλοντα Natura 2000. Δεν δικαιολογείται επομένως ούτε από τα στοιχεία τα συγκεκριμένα, ούτε από την ενδεχόμενη επίπτωση του ε, ξενοδοχειακού αυτού συγκροτήματος. Δεν υπάρχει επίπτωση ε, από την οικοδόμηση του ε, συγκροτήματος ή στο περιβάλλον. Βεβαίως, εάν η Κομισιόν έχει κάποια άλλα στοιχεία θα πρέπει να μας τα πει. Ευχαριστώ πολύ Φερνάντο. Καλό είναι να δίνουμε το λόγο σε κάποιον, αλλά ακόμα καλύτερο είναι όταν μας τον επιστρέφουν. Ωραία, το λόγο τώρα έχει η Άγγελα και παρακαλώ να είστε σύντομοι γιατί πρέπει 12 και μισή ακριβώς να σταματήσουμε. Μην επαναλαμβάνεστε γιατί λέτε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Θα προσπαθήσω εγώ, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να θυμίσω και το λέω στον Χουαν Φερνάντο και το λέω και στην Κομισιόνα. Εάν ζητούσαμε, ε, αν ζητήσαμε ε, να συζητήσουμε το θέμα αυτό το θέμα αυτό να το δούμε επιγόντως λέω είναι γιατί ε, είχε αρχίσει μετακίνηση εδαφών χωρίς πρώτερη αδειοδότηση. Ε, τα έργα ξεκινούν με την αδειοδότηση ε, και ακριβώς γι' αυτό ζητήσαμε, γι αυτό ζητήσαμε την επίγουσα διαδικασία γιατί είχαν ξεκινήσει έργα. Ε, στην, όπως ε, είπαν και οι αναφέρουσες ε, έχουν ήδη συλλεγεί πάνω από 100.000 υπογραφές κατά αυτού του, αυτής της οικοδόμησης, κατά αυτού του ξενοδοχείου. Έχουν γίνει διαβουλεύσεις και επομένως θα πρέπει να μελετήσουμε εάν και κατά πόσον έχουν καλυφθεί οι περιβαλλοντικές υποχρεώσεις. Όχι, εδώ βλέπουμε βλέπουμε ότι ε, αυτή η παραλία της Λατεχίδα είναι ακριβώς δίπλα, άπτεται ε, της προστατευόμενης περιοχής της Μοντάνια Ρόχα ε, και επομένως ε, δεν είναι δυνατόν να το ξεχάσουμε αυτό επίσης να σας πω ότι το 1994 έχει ε, ζητήσει ακριβώς ε, το ε, έχει ζητήσει να δημιουργηθεί μια, ειδική, μια ζώνη ειδική συντήρησης που συμπεριλαμβάνει και την παραλία της Λατεχίδα και βεβαίως το γειτονικό μοντάνια, τη γειτονική μοντάνια Ρόχα και επομένως δεν είναι δυνατόν εδώ να επιτραπεί η οικοδόμηση ενός τέτοιου ξενοδοχείου βεβαίως δεν μπορούμε να σταματήσουμε την ανάπτυξη ή δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε την την, ε, ε, ε, την ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να προλάβουμε γιατί αν προκύψει ζημία αυτή η ζημία θα είναι πλέον χωρίς επιστροφή. να προλάβουμε λοιπόν πριν έχουμε μπροστά μας την καταστροφή. Τον Ιανουάριο, ε, τον προηγούμενο, ήδη εγώ είχα ε, υποβάλει σχετικό αίτημα στον ε, Επίτροπο, ο οποίος απήντησε ότι είμαι βέβαιος ότι οι ισπανικές και τοπικές αρχές θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να υπάρξει ε, ε, συμμόρφωση ε, με την οδηγία Natura 2000. Αλλά ήδη ξεκίνησαν τα έργα, ήδη άργησαν οι εξκαφές και επομένως θα πρέπει να το δούμε γιατί όντως η τοπική κυβέρνηση και η ισπανική κυβέρνηση είναι αυτή. Τώρα το έχω εμπιστοσύνη ότι η κυβέρνηση θα πάρει τα απαραίτητα. Όχι, δεν σημαίνει τίποτα το έχω εμπιστοσύνη. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη, ελέγχουμε εάν υπάρχει συμμόρφωση με τους νόμους. Γι' αυτό λοιπόν εγώ για μία ακόμα φορά λέω ότι θα πρέπει να ε, δούμε και να εφαρμόσουμε την αρχή της ε, πρόληψης και η Κομισιόν θα πρέπει να απαντήσει από αυτού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Πρώτα απ' όλα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ότι από τη στιγμή που μιλάμε για μια περιοχή η οποία βρίσκεται δίπλα ε, σε προστατευμένη ζώνη και δίπλα πάλι και συνορεύει ε, με το δίκτυο Natura, οπωσδήποτε οποιαδήποτε κίνηση και οποιαδήποτε δόμηση ε, τις προστατευμένες αυτές περιοχές τις, τις επηρεάζει. Και εδώ μιλάμε για οικοδόμηση ακριβώς στα όρια αυτών των προστατευμένων ε, περιοχών. Γιατί διαφορετικά και αν δεν ε, κινηθούμε τώρα, όπως είπε και η Άγχελα προηγουμένως, ε, θα είναι πολύ αργά όταν θα καταλάβουμε ότι κάτι τρέχει. Τώρα το γιατί δεν μας ενδιαφέρει όταν θα έχουν γίνει οι παράνομες κατασκευές να διαπιστώσουμε την παρανομία. Και το λέω γιατί ε, ε, εγώ έρχομαι, είμαι από τη Βαλένθια και είδαμε ε, τέτοια διαδικασία κοντά στο λιμάνι και είδαμε ακριβώς ότι εκ των υστέρων διαπιστώσαμε «Α, ναι, τόσα χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα τα οποία παράνομα έχουν χτιστεί». Εδώ μιλάμε οπωσδήποτε για μία αδειοδοτημένη κατασκευή με άδεια οικοδόμησης η οποία όμως βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην προστατευμένη παραλία Λατεχίδα και δίπλα στην ε, προστατευμένη περιοχή της Μοντάνια Ρόχα. Δεν είναι δυνατόν για μία ακόμα φορά ε, εκ των υστέρων και όταν όλα θα έχουν γίνει να πούμε «Α, ναι, συνέβη το αναπόφευκτο». Ευχαριστώ πολύ, κύριος Καλμή. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι που επιτέλους ένα ισπανικό θέμα έρχεται σε αυτή την Επιτροπή. Ε, ε, εδώ και καιρό δεν είχαμε δει ισπανικό θέμα. Χαίρομαι λοιπόν. Εάν φύγει η Ισπανία, η Επιτροπή μας θα μείνει χωρίς δουλειά. Εγώ θα πω κάτι απλό. Ενστερνίζομαι τα όσα είπε η Κομισιόν. Μη ζηλεύετε, μη ζηλεύετε και η Γερμανία πολλές αναφορές έχει. Τώρα, του, ο συνάδελφος Λόπες Αγγελιάρ είπε πολλά σωστά πράγματα ε, και μη λησμονούμε ότι η πολιτική είναι οπωσδήποτε και η, και η διακυβέρνηση μάλλον είναι ε, η ε, πολιτική των ισορροπιών. Τα ξέρουμε όλα αυτά, έχουμε, γνωρίζουμε την περιοχή Δεν θέλουμε τώρα να δούμε, τι έγινε παλιά, αλλά ε, ε ένας, ε, ένας δικηγόρος ε, είπε να πας με τον νόμο και ο άλλος δικηγόρος είπε αμήν. Okay, um, now we are about to conclude, but I would... Εντάξει, φτάνουμε στο τέλος του κατάλογου, κατάλογου μιλητών. Να δώσουμε το λόγο στην αναφέρουσα για δύο λεπτά το πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, νομίζουμε ότι η, τα εκατομμύρια των Ευρωπαίων πολιτών ε, τουριστών που έρχονται Πιστεύουμε ότι έρχονται γιατί ακριβώς ε, εκτιμούν ε, και το ε, περιβάλλον μας. Ε, ξέρετε, εν, πριν από έναν αιώνα περίπου, ο Λεόν Θεοροδρίγες, ο ποιητής μας είπε ότι εάν ξεγυμνώσουμε από τις ομορφιές του, την, από τις ομορφιές της τη γη μας, τότε δεν θα μείνει τίποτα ούτε από την ομορφιά, ούτε από τις πηγές της υγείας. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα προβλήματα και όσον αφορά τα της αποχετεύσεις. Ήδη ε, έχουμε πρόβλημα όσον αφορά την μη συμμόρφωση ε, με την ε, οδηγία πλαίσιο για, την, για το βιολογικό καθαρισμό των υδάτων κλπ. Ε, υπήρξε πριν από χρόνια μία ε, αναφορά ε, η οποία αναφέρει ότι στην κύρια περιοχή η οποία είναι πάρα πολύ κοντά στην παραλία ε, έχουν διαπιστωθεί ιδιαίτερα προβλήματα όσον αφορά στάσιμα νερά, όσον αφορά ε, ε, νερά τα οποία προκαλούν, δημιουργούν έλλη που μυρίζουν άσχημα και τα οποία είναι ακριβώς νερά τα οποία προκύπτουν, φτάνουν μέχρι την παραλία ακριβώς από τις αποχετεύσεις των σπιτιών. Δεν είναι όμβρια ύδατα ή πρόκειται ακριβώς για τις αποχετεύσεις ε, των ε, σπιτιών και των ε, δομημένων περιοχών που φτάνουν μέχρι αυτή την παραλία. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν σε ένα πρόβλημα το οποίο ήδη υπάρχει και σε μια μη συμμόρφωση η οποία είναι ήδη διαπιστωμένη να προσθεθεί και το, το πρόβλημα των αποχετεύσεων αυτού του συγκεκριμένου ξενοδοχείου. Πρόκειται επομένως και για θέμα υγείας της περιοχής. Επίσης, να σας πω ότι εκτός από την άδεια για αυτό το ξενοδοχείο έχει ε, άδεια ο ίδιος οικονομικός όμιλος για την οικοδόμηση 40 bungalows ε, τα οποία θα είναι και αυτά δίπλα σε αυτήν την παραλία την οποία προσπαθούμε να σώσουμε. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ και για τον ενθουσιασμό σας, τον χρόνο σας, ε, τις προσπάθειές σας. Αν ο κόσμος ε, ήταν γεμάτος ανθρώπους σαν και εσάς, θα ήταν ένας πολύ καλύτερος τόπος. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την ανασχόλησή σας, αλλά και για το γεγονός ότι ταξιδέψατε μέχρι τις Βρυξέλλες, παρότι προέρχεστε από τα Καναρέ από την Τενερίφη και ήρθατε σήμερα στις Βρυξέλλες, κατανοώ ότι είναι μεγάλη θυσία για σας. Σας ευχαριστώ όμως για αυτή τη θυσία που κάνατε για τον ε, σκοπό για τον οποίο πολεμάτε. Σας ευχαριστώ εγώ όλους, λέει μιλήτρια Κλείνουμε αυτό το σημείο. Και αν συμφωνείτε, να κάνουμε το εξή. Ξέρετε ότι το άρθρο 6 της Οδηγίας Οικοσυστημάτων εφαρμόζεται εδώ και κάθε αναπτυξιακό έργο θα πρέπει, ή κατασκευαστικό έργο θα πρέπει να συμμορφούνται με αυτόν τον κανόνα. Αυτό αναμφίβολα. Επομένω, μπορούμε κατεπηγόντως να στείλουμε επιστολή αύριο τις τοπικές, περιφερειακές αλλά και εθνικές αρχές στην Ισπανία να ζητήσουμε ξεκάθαρα μία αξιολόγηση αντικτύπου. Από ό,τι φαίνεται δεν έχει γίνει. Και αν όχι, τότε δεν υπάρχει πλήρη συμμόρφωση με το άρθρο 6 της Οδηγίας Περικοσυστημάτων που απαιτεί πριν από οποιαδήποτε κατασκευή να γίνει ε, πλήρης αξιολόγηση αντικτύπου. Όπως έχουν αναφέρει συνάδελφοι προηγουμένω, αλλά και εσεί. αυτή η κατασκευή ενδέχεται να οδηγήσει σε μία αναστρέψιμη ζημιά για το περιβάλλον. Και εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να λαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Γι' αυτό βρισκόμαστε στον πλανήτη, γι' αυτό βρισκόμαστε κάποιοι από εμά εδώ στο Κοινοβούλιο. Αυτή είναι μια πιθανή διέξοδος λοιπόν. Και βέβαια η Γραμματεία θα βρίσκεται συνεχώ σε επαφή με την Επιτροπή για αυτό το ζήτημα για να δούμε πώ θα προχωρήσουμε. Παραμένει ανοιχτή όμω η αναφορά. Θα κάνουμε αυτέ τι κινήσει. Συμφωνούν οι συνάδελφοι. Ωραία. Ευχαριστώ. Ευχαριστημένε και οι αναφέρουσε. Το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα λοιπόν. Σα ευχαριστώ. Καλό διάλειμμα και τα λέμε το απόγευμα.